Yes, friends. Καλημέρα ε, φίλοι, ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Ε, καλώς ήρθατε στην ε, συνάντηση που θα διαρκέσει ολόκληρη την ημέρα. αρχικά θα κινηθούμε με βάση την ημερήσια διάταξη. Ας περάσουμε αρχικά στις ανακοινώσεις. Υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από φινλανδικά, ε, κροατικά και βουλγαρικά. Επίσης θα έχουμε ομάδες επισκεπτών στις 25 Απριλίου, σήμερα δηλαδή. Ο κύριος Μπροκ ε, κάλεσε 30 επισκέπτες ε, από το Belgian Youth Diplomacy που θα έρθουν αργότερα και οι ευρωβουλευτές ε, Κάρη και Λόπες ε, προσκάλεσαν από την ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές σχετικά ε, για σήμερα για να παρακολουθήσουν την ε, ψηφοφορία σχετικά με, το, με την ε, δέσμη οδικής μετακίνησης. Επίσης υπάρχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο από την κυρία Μωρίν σχετικά με την ψηφοφορία για την οδηγία της απόσπασης εργοζομένων ενώ επίσης υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα της Επιτροπής η συνάντηση της 16ης και 17ης Μαΐου μεταφέρθηκε για τις 14 ε, και 15 Μαΐου Σύμφωνα λοιπόν με την καινούργια ε, ημερήσια διάταξη, μισό λεπτό να σας δώσω τα ακριβή στοιχεία, ε, από τις 3 με 6.30 την ε, Δευτέρα 14 Μαΐου και στη συνέχεια την Τρίτη 15 Μαΐου από τις 9 με 12.30 και στη συνέχεια από τις 2.30 μέχρι τις 6.30. Ε, Σχετικά με το σημείο 5 θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα υπάρξει ε, μια έκτακτη συνάντηση στις 24 Μαΐου όπου θα ε, γίνει ανταλλαγή απόψεων ε, με τον Επίτροπο Τροπρόφσκι ε, και θα έχουμε επίσης την Επίτροπο Τάισεν σχετικά με μια πρόταση που έχει γίνει για την ΕΛΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ύστερα από απόφαση συντονιστών στις 15 Μαΐου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ψηφοφορία στον διαρθρωμένο διάλογο και ένα εργαστήριο πάνω στο ε, θέμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Αυτές ήταν όλες και όλες οι ανακοινώσεις, ε, η έγκριση των ε, πρακτικών της 21ης και 2ης Μαρτίου. Ο κύριος Μπέκερ. Καλημέρα, ε, Πρόεδρε. Ε, έχω ένα μικρό αίτημα. Ε, μία απάντηση σχετικά με το ερώτημά μας. Θα μπορούσατε να επιβιώσατε ότι το καποτάζ θα συμπεριληφθεί στη σημερινή ψηφοφορία. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, θα συμπεριληφθεί. Και θα περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης ε, σχετικά με το σχέδιο οικονομισμού για τις κοινωνικές στατιστικές. Ε, το οποίο επεξεργαζόμαστε στις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τον κανονισμό για τις κοινωνικές ε, στατιστικές. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Μέστσερης. Ε, η συζήτηση έγινε στις 27 Μαρτίου και οι συνομοθέτες ε, παρουσίασαν τις θέσεις τους και συμφώνησαν πάνω σε ένα ε, πρόγραμμα εργασίας. Ε, έγιναν συνολικά τρεις συναντήσεις σε τεχνικό, σε τεχνικό επίπεδο, ενώ ο, τρίτο, ο δεύτερος τριμερής διάλογος θα γίνει αύριο, ενώ η επόμενη αναφορά σχετικά αφορά τις υπηρεσίες υπό την Επιτροπή η συνάντηση έγινε χθε και μαζί με μένα ε, το Κοινοβούλιο εκπροσωπούνταν από τον κύριο Σοντέλ, ο οποίος είναι εισηγητής για την ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ε, είχαμε εκπρόσωπο από το υπεύθυνο για το Eurofund ε, και το ΩΣΑ και αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε διάφορα θέματα ε, τα οποία συζητηθούν στις 22 Μαΐου, τα οποία δεν προλάβαμε να επεξεργαστούμε ε, χθες ε, λόγω των έντονων συζητήσεων που είχαμε για διάφορα άλλα θέματα. Ε, προσδοκούμε να υπάρξει περαιτέρω ε, πρόοδος ε, σε τεχνητικό επίπεδο για τη συνάντηση της 22 Μαΐου. Αυτές ήταν οι εκθέσεις και περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που αφορά το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιδοτικό προϊόν και το λόγο έχει ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι η ε, συγκεκριμένη έκθεση η οποία συζητείται σε συνολικά τρεις ε, επιτροπές ε, της ΕΚΟ, και ΕΜΠΛ μπορώ να σας πω αρχικά ότι έχουμε επικοδομητικούς διαλόγους μεταξύ των εισηγητών και των τριών επιτροπών και σε πολλούς τομείς ε, μπορούμε να βρούμε μια ε, συμφωνία, μια ευρεία συμφωνία. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ωστόσο ε, και θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω την πορεία η οποία αφορά την δική μας Επιτροπή. Αρχικά θα ήθελα να τονίσω ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής ε, ώστε να εξελίξει το συγκεκριμένο προϊόν ε, θα θέλω να το χαρακτηρίσω ως κάτι αξιέπαινο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ε, βήμα προς την ευρωπαϊκή κοινωνική εξέλιξη και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα ξεκάθαρα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Τώρα ποιος είναι ο στόχος μας. Υπάρχουν διάφορες προτεραιότητες. Μία εξ αυτών είναι ότι ε, το ΠΕΠ θα πρέπει ε, να είναι ένα μακροπρόθεσμο προϊόν αποταμίευσης ε, διότι κυρίως αφορά για ένα ελκυστικό προϊόν για την σύνταξη. Το ΠΕΠ, το ΠΕΠ στοχεύει κυρίως τους νέους που θα τους διασφαλίσει μια σιγουριά στα γεράματα θα πρέπει να είναι διαφανές και, να, και διασυνοριακό και θα ήθελα να τονίσω ότι ο πανευρωπαϊκός χαρακτήρας ε, θα πρέπει να είναι μια υποχρέωση την οποία θα πρέπει να τηρήσει το Κοινοβούλιο στην τελική έκθεση όλων των επιτροπών διότι είμαστε πεπισμένοι ότι οι πάροχοι ε, ΠΕΠ μπορούν να φροντίσουν και οφείλουν να φροντίσουν ε, με τις ε, συνεργασίες και τις εταιρικέ τους σχέσεις ε, στις διάφορες χώρες να δημιουργήσουν μια πανευρωπαϊκή παρουσία ακόμα και αν δεν έχουν κάποιο υποκατάστημα σε άλλη χώρα. Ο πανευρωπαϊκός λοιπόν χαρακτήρας για μένα είναι υψής της σημασίας. Ε, αυτό το είδος ε, ευρωπαϊκής ασφάλειας κεφαλαίου ε, σίγουρα θα προσεγγιστεί πιο συγκεκριμένα στις συζητήσεις του Κοινοβουλίου και είμαι πεπισμένος ότι εδώ πέρα θα έχουμε ένα μοναδικό προϊόν σε περίπτωση που έχουμε ένα κεφάλαιο ε, ένα ε, ε, κεφαλαιακό κεφάλαιο για όλη την Ευρώπη. Ε, πιστεύω ότι ε, ο πανευρωπαϊκός χαρακτήρας είναι ύψης της σημασίας λοιπόν. τώρα κάθε χώρα θα πρέπει να συμμετέχει στο ΠΕΠ ε, διότι θεωρούμε ότι για εκατομμύρια Ευρωπαίους ε, πολίτες ε, θα μπορέσει να δώσει δυνατότητα σε πολίτες όπου ζουν σε χώρες όπου δεν υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες, για παράδειγμα αρκετές ανατολικές Ευρωπαϊκές και νοτιοευρωπαϊκές χώρες ε, σε αντίθεση με χώρες οι οποίες έχουν πιο ανεπτυγμένα κοινωνικά συστήματα. Εκεί λοιπόν το ΠΕΠ θα μπορεί ε, να είναι μια επιπλέον διασφάλιση ε, της ποιότητας διαβίωσης στα γεράματα. Το ε, ΠΕΠ ε, λοιπόν θα ήταν ένα τρομερό δώρο ε, για τους, από τους μεγάλους προς τα παιδιά τα οποία στην συνέχεια θα μπορούν να αποπληρώνουν τα συγκεκριμένα συμβόλαια. Όσον αφορά την απόδοση του ΠΕΠ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε το EPRS για την ενημέρωση. Η αξιολόγηση αυτή συμπεριλαμβάνεται σε κάθε έγγραφο το οποίο σας έχω ε, καταθέσει και δείχνει ε, σε μία, ε, σε μία απόδοση της τάξεως του 4% για 40 χρόνια αν ε, δούμε τα τελευταία 40 χρόνια, τότε θα δούμε ότι δεν απέχουμε ε, πολύ. Αν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ένας νέος άνθρωπος ε, πληρώνει για 40 χρόνια και στη συνέχεια φτάνει τα 40.000 ευρώ, τότε αναγνωρίζουμε ότι με όλα τα μοντέλα υπολογισμού, τα οποία δεν έχουν πολύ υψηλά κόστη παροχής και συμβολή, συμβουλέου αναγνωρίζουμε ένα ε, μοντέλο ε, το οποίο ε, παρουσιάζει μια πολύ ικανοποιητική εξέλιξη του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, στο κόστος της τάξης του 1,5% και 40.000 ευρώ ε, ε, συνολικές καταθέσεις έχουμε συνολικά 44.000 ευρώ στο οποίο συνυπολογίζεται το 4% πληθωρισμός. Οπότε είμαι βέβαιος κάτι το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό δεν θα μπορούσα να σας το υποσχεθώ. αυτά είχα λοιπόν ε, να πω. Ε, θα ήθελα να τονίσω και κάποια άλλα, ε, άλλες μικρές λεπτομέρειες. Ε, βλέπουμε την ποιότητα ε, του ε, ΠΕΠ στο να κλείσει το χάσμα ε, της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των φύλων. Βλέπουμε λοιπόν γυναίκες οι οποίες ακολουθούν μια καριέρα και οι οποίες θα προσελκυθούν ιδιαίτερα από το ΠΕΠ. Ξεκαθάρισα το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα ε, του ΠΕΠ και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ε, επικουρικό ε, πρόγραμμα είναι ξεκάθαρο, όμως για πολλούς ίσως να μην είναι επικουρικό, αλλά να είναι η μόνη ε, συνταξιοδοτική πρόνοια που θα έχουν Τώρα όσον αφορά το ζήτημα της φορολόγησης θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι εδώ δεν έχουμε καμία επιρροή ε, δεν μπορούμε αυτό το ε, ερώτημα να το ε, χειριστούμε διότι δεν υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το θέμα ε, θα το ζητήσουμε αυτό και θα το ξεκαθαρίσουμε και κατά την άποψή μου ε, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό ούτω ώστε ε, κάθε κράτος μέλος να προσφέρει φορολογικά ωφέλη στο ΠΕΠ όπως προσφέρονται και σε άλλα προϊόντα εξοικονόμησης. Ε, λέμε ε, λοιπόν την ε, πιο φιλική προσέγγιση από φορολογικής άποψης όσον αφορά το ΠΕΠ. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κόστη εάν ένας πάροχος δεν είναι παρόν σε ένα κράτος μέλος. Δεν, θα, δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν το πώς θα μπορεί να είναι κάποιος ε, παρόν σε κάθε κράτος μέλος μπορεί να υπάρξει εταιρική ε, σχέση. Ε, τα κόστη είναι μια δύσκολη συζήτηση. Περιμένουμε από τους παραόχους να είναι δίκαιοι και να λαμβάνουν το κοινωνικό στοιχείο υπόψη τους και το ένα ανώτατο όριο του 5% ε, είναι αυτό το οποίο, στο οποίο κινούμαστε. Ε, μπορώ να φανταστώ ότι η διαφάνεια του ε, ΠΕΠ θα πρέπει να είναι τόσο ξεκάθαρη και καλά οργανωμένη, ούτως ώστε η πάροχοι ε, ΠΕΠ Ε, να κάνουν τα προϊόντα τους τον τελευταίο 20 χρόνων ε, διαφανή, για ποιο λόγο 20 και όχι 5, θέλουμε όλο το χρονικό πλαίσιο και πριν την χρηματοπιστωτική κρίση του 8 να συμπεριληφθεί. Ε, και αυτό θα βοηθήσει τους πολίτες να καταλάβουν πως ένα συνταξιοδοτικό προϊόν κινήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση. Ε, και όσον αφορά τις, ε, τους ε, παράγοντες υπάρχει η λεγόμενη default option, ένα σταθερό προϊόν. Πιστεύω ότι η Κοινωνική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τουλάχιστον ένα από τα ε, παρεχόμενα προϊόντα να είναι ένα τέτοιο ε, προϊόν default ε, και να περιλαμβάνει όλη την ποιότητα της διασφάλισης κεφαλαίου. Αν τώρα υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία με διαφορετικούς φακέλους θα μπορούν να παρασκευθούν, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ δεν θέλω να το αποτρέψω, όμως σίγουρα ένα εξ αυτών θα πρέπει να έχει αυτή την εναλλακτική default. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, ε, στην επόμενη φάση θα ήθελα να σας ζητήσω να ολοκληρώσετε τις ε, τρομπολογίες. Ε, η επόμενη εβδομάδα, 2 Μαΐου, μέχρι τότε μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε αυτήν την καλή συνεργασία και με τους σκιώδεις. Ε, και στις 28 Ιουνίου θεωρώ ότι ε, θα ε, μπορούμε να έχουμε μια καλή, ένα καλό αποτέλεσμα για την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ για αυτήν την εισαγωγή. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, σκιώδες, ε, σκιώδες αρχικά η κυρία Ρένα, από ε, η κυρία Ιγγέριος αντικαθιστά την κυρία Ρένα. Δεν την αντικαθιστώ ακριβώς. Η Μαρία Ρένα λείπει σε αποστολή. Και εμείς εξακολουθούμε να συζητούμε στην ομάδα εργασίας μας την θέση μας απέναντι στο ΠΕΠΑ. Είναι καλό πάντως που αν μη τι άλλο αυτό που μπορώ να πω σαν πρώτη αντίδραση σε αυτά που μας είπατε είναι ότι ναι, είμαστε θετικά. Αντιμετωπίζουμε θετικά το ζήτημα αυτό γιατί πιστεύουμε ότι όντως θα καλύψει το σταξιδωτικό κενό για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε. Κυρίως όσον αφορά τους πιο ηλικιωμένους και βλέπουμε στην Ευρώπη ότι έχουμε όλο και περισσότερους ηλικιωμένους. Οπότε επήγει να βρεθεί μια λύση για να καλυφθεί το κενό αυτό. Τώρα, πιο συγκεκριμένα. Επί της αρχής, πρέπει να σκεφτούμε πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Ένα συνταξιδιωτικό πρόγραμμα πρέπει να διατίθεται για τον κόσμο και πρέπει να προσφέρει κατάλληλες συντάξεις. Όμως, ανάμεσα στα όνειρα και στις πράξεις υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν αρχές, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Και μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι ανάμεσα σε αυτά τα δύο τα εμπόδια είναι τεράστια. Προκειμένου λοιπόν να εξετάσουμε την πρόταση αυτή, προσπαθούμε να δούμε το ΠΕΠ, αυτό δηλαδή το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Σταξιδιωτικό Προϊόν, σαν συμπλήρωμα ώστε να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν μια ικανοποιητική σύνταξη. Θα πρέπει δηλαδή να αποτελεί προσθήκη και να μην αντικαθιστά τις ε, κατάλληλες συντάξεις του πρώτου δεύτερου πυλώνα. Για τελειώς πάμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Οπότε για μένα, και βέβαια μιλάω εξ ονοματός μου και δεν μιλάω εντελώς εκ μέρους της ομάδας μου, νομίζω ότι θα ήταν καλό να είχαμε μια καλή διατύπωση στις αιτιολογικές σκέψεις, μια σαφή διατύπωση που να λέμε αυτό είναι που θέλουμε, αυτός είναι ο στόχος μας με την πρόταση αυτή, να πρόκειται για προσθήκη και να μην αντικαθιστά κανένα άλλο σταξιδωτικό πρόγραμμα. Ίσως θα μπορούσαμε επίσης να το διατυπώσουμε κι αλλιώς, να πούμε ότι μετά από πέντε χρόνια να δούμε κατά πόσο πράγματι λειτουργεί σαν πρόσθετη σύνταξη για τις νέες γυναίκες, για παράδειγμα, αν αρχίζουν ένα πέψ σαν συμπλήρωμα ή όχι, αν είναι οι αυτοπασχολούμενοι περισσότερο που χρησιμοποιούν ε, το μηχανισμό αυτό του ΠΕΠΣ για να έχουν μια ικανοποιητική σύνταξη αργότερα. Πρέπει να είναι σαφής λοιπόν ο στόχος μας και να αποτελέσει μέρος της πρότασης ότι θα ξαναδούμε μετά από κάποια χρόνια κατά πόσο αυτή η πρόταση πραγματικά λειτουργεί σαν ε, προσθήκη ή τελικά αντικαθιστά τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Γκέρι και έπρεπε να είναι εδώ η κυρία Μακιντάιρ τον αντικαθιστά όμως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα το πρωί ο κύριος και γι' αυτό θα σας μεταφέρω την άποψη της ομάδας μου του ΙΣΙΑΡ. Πρώτα απ' όλα θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέκερ για την γνωμοδότησή του αυτή. Χαίρομαι πολύ για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχει συμπεριλάβει. Και σίγουρα θα στηρίξουμε το κείμενο. Κάποια πράγματα με χαροποιούν όλος ιδιαίτερος, όπως η ενίσχυση αυτής της εθελοντικής επιλογής. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό στοιχείο. Έπειτα πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος αυτό για την ε, σύνταξή του, ότι πρόκειται για τα γερατιά του. Και το θέμα αυτό της μεταφοράς διασυνοριακά των ε, συντάξεων είναι πολύ θετικό. Οπότε όλα αυτά πολύ μου αρέσουν. Στην ε, τροπολογία 9 λέμε ότι πρόκειται για ένα νέο συμπληρωματικό μέσο στα ήδη υπάρχοντα εξωτερικά προγράμματα. Αυτό για μας είναι στοιχείο κλειδί. Αυτό το οποίο μας απασχολεί όμως περισσότερο και μας ανησυχεί είναι το θέμα της φορολόγησης. Δεν θέλουμε να στηρίξουμε καμία ιδέα φορολογικής αναρμόνισης και στην παρουσίαση του κύριου Μπέκερ αναγνώρισε ότι το φορολογικό είναι εκτός πεδίου εφαρμογής, ε, δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πράγματι δεν είναι κάτι που εμπίπτει στις αρμοδιότητες τη δικιάς μα επιτροπή, όπω και να έχει το πράγμα. Αλλά ήθελα να το έχω πει ότι είναι μια ανησυχία μα αυτό, η φορολόγηση. Πάντω σα ευχαριστώ πολύ για το έργο σα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά αυτή και πρέπει όλοι να ενθαρρυνθούν στην Ευρώπη να έχουν το δικό του ατομικό σταξιδωτικό προϊόν. Έχουμε συζητήσει για τον πυλώνα 1, 2 και 3 και κατά το παρελθόν. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά. Αλλά αυτό που δεν θέλω είναι η περιπλοκότητα όλων αυτών των ζητημάτων των πυλώνων να έρθει και να μπει μέσα σε αυτό το πανευρωπαϊκό ατομικό σταξιδιωτικό προϊόν, το οποίο είναι αναγκαίο και δεν θέλω να προκύψουν τέτοιες δυσκολίες. Πάντως, ευχαριστώ πολύ τον Χαντσπέκερ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Καλβεσαμπό από την Άλντε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω ισπανικά. Η ομάδα μου, Άλντε, καλωσορίζει και με ιδιαίτερη ικανοποίηση αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία αυτή, αυτή την πρόταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κύριοι Ντομπρόσκε και Καϊτάνεν, γιατί δεν είναι το Μοσκοβισί ούτε υπεύθυνο για την απασχόληση, έχουν μια γενική έτσι, άποψη των ε, προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη φτώχεια ας πούμε, στην Ευρώπη και προσπαθούν να βρούνε λύσεις, πρακτικές λύσεις. Απτές και ευρωπαϊκές. Κάτι το οποίο σήμερα που λείπει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι καλό νέο. Για μας λοιπόν είναι περισσότερο που ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή, είναι καλή και θα τη στηρίξουμε καταρχήν, έτσι. Γιατί θέλουμε να υλοποιηθεί, θέλουμε να προχωρήσει στο Συμβούλιο, ναι. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει εμπόδια η Άλντε. Όμως, κατόπιν τούτων, η Άλντε χαίρεται πολύ και με τη δουλειά του κύριου Μπέκερ που είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης πιστεύουμε ιδιαίτερα θετικό. Επικεντρώνεται πραγματικά στα προβλήματα τα οποία πρέπει να εξετάζει η Επιτροπή Απασχόλησης και που είναι η προστασία των πολιτών, των μελλοντικών συντοξιούχων και να διασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς από τη μία χώρα στην άλλη τη σύνταξη, την ενημέρωση την καλή, τη διαφάνεια για τα συνταξιδοτικά την ασφάλεια, για την Ευρώπη αυτό καλείται να προσφέρει. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συσσόρευση και την αποσυσσόρευση. Τα διάφορα στάδια αυτά να μην κοστίζουν χρήματα στον ε, αποταμιευτή. Να υπάρχει καλή ενημέρωση στους χρήστες. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν λοιπόν στη συνέχεια, δεν θα μπούμε τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να λυθεί. Υπάρχουν τα άρθρα 23 και 34 που θα ήθελα να συζητήσουμε με τον εισηγητή. Η Άλντε μπορεί να έχει και την τύχη ο εισηγητής στην ΕΚΟ που είναι η κυρία Σόφι Φαντεβέλτ προέρχεται από την ομάδα μας, από την Άλντε και έτσι βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή μαζί της. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ε, εν πάση περιπτώσει, ώστε να βγει κάτι όσο γίνεται καλύτερο κοινωνικά και οικονομικά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, εκτός από μία ίσως, που πιστεύω ότι είναι σημαντική για την ομάδα μου. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό προϊόν, έτσι, ευρωπαϊκό. Και αφού πρόκειται για κάτι που θα δημιουργήσουμε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, τον έλεγχο αυτού του νέου προϊόντος, την επίλυση διαφορών που ενδεχομένω θα προκύψουν, την εποπτεία θα την έχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, που ήδη υπάρχει αυτή η αρχή, έτσι. Δεν πρέπει ούτε να επαναθνικοποιήσουμε κάτι, ούτε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Γι' αυτό το λέμε ευθύ εξ αρχή, γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα επίμαχο ζήτημα, δεν ξέρω. Οπότε ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπάκερ για το εξαίρετο έργο του. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στις απόλυτα θεμητές επιθυμίες όλων. Αλλά καταρχήν λέμε ότι συμφωνούμε πως είναι ένα καλό προϊόν, μπορεί να βελτιωθεί και πρέπει να προστατεύονται καλά οι χρήστες. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. προεδρο ευχαριστούμε. Περνάμε στην ΚΟΕ. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι εδώ ή την αντικαθιστά κάποιος. Α, εδώ είσαστε βεβαίως, βεβαίως, συγγνώμη. Συνήθως κάθεστε από την άλλη μεριά, γι' αυτό μπερδεύτηκα και δεν σας εντόπισα μέσω. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Συνήθως εγώ κάθομαι πιο δίπλα στην πόρτα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την περασμένη Παρασκευή το Προεδρείο της ομάδας μου, η Γκουέντζιελ, επισκέφτηκε τη Σόφια, όπου και πραγματοποίησε μια ειδική συνεδρίαση. Σε αυτήν τη συνεδρία συμμετείχαν πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, μη και συνδικαλιστές. Γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί με τρόμο, ναι δεν το υπερβάλλω, ακούσαμε ένα από επίσημα χείλη ότι σχεδόν ένας στους δύο συνταξιούχους, για την ακρίβεια το 46% των συνταξιούχων, λαμβάνει μια σύνταξη που δεν ξεπερνά 164 ευρώ. 164 ευρώ και θεωρείται καλή σύνταξη γιατί η χαμηλότερη είναι γύρω σε 100-110 ευρώ. Αλλά και στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί μέσα σε μια επταετία πάνω από 25 μειώσεις στις συντάξεις τους. Και αν κοιτάξουμε σε ακόμη μια γειτονική χώρα, τη Ρουμανία, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Την ίδια ώρα, ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες οι δημόσιες συντάξεις έχουν πάρει την κατιούσα. Επομένως, σε ποιον επευθύνεται αυτή η δημοτική, ιδιωτική σύνταξη την οποία συζητάμε σήμερα, υποτέθω στους πλουσιότερους που μπορούν να την αγοράσουν. Δηλαδή, σε αυτούς που έχουν καταθέσεις και επειδή δεν θέλουν να αγοράσουν μετοχές στο χρηματιστήριο, γιατί θυμούνται τη χρηματοπιστωτική πιστοτητική κρίση το 2008 και θέλουν κάτι πιο ασφαλές. Πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο δώρο στις τράπεζες και στις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο. Άλλωστε, η έκθεση της Κομισιόν είναι σαφής. Θέλει να μεταφέρει χρήματα από τις καταθέσεις της κεφαλαίας Έτσι θα υπολογίσουμε την αρχή των κοινωνικού πυλώνα για βιώσιμα συντάξεις με την πανευρωπαϊκή ιδιωτική σύνταξη και για ποιους λόγους. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία με την οποία σχεδόν διαφημίζεται η ιδιωτική σύνταξη ως το σημαντικότερο υποκατάστατο για τον δεύτερο πυλώνα συντάξεων δημιουργεί πολλούς κινδύνους για το δημόσιο σύστημα συντάξεων τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα καθώς και για τις επαγγελματικές συντάξεις. Και αυτούς τους κίνδυνους θα αναδείξουμε και με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από τους πράσινους. Η Τζιν Λάμπερτ δεν είναι όμως εδώ ότι να αντικαθιστά κανείς. Όχι, κανείς από τους πράσινους. Η FTD. Είναι εδώ κανείς. Όχι. Όχι, δεν βλέπω κανέναν. Η ΕΝΕΦ. Εδώ. Είστε εδώ κύριε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όντω, πολλά ερωτηματικά θέτει η υπόθεση αυτή, γιατί πρόκειται για μια ρύθμιση για ένα πανευρωπαϊκό προϊόν ε, συνταξιδοτικό, το οποίο δεν αποτελεί ούτε υποχρεωτική βασική σύνταξη, ούτε συμπληρωματική υποχρεωτική, ούτε εθελοντική συμπληρωματική των εθνικών καθεστώτων. Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό προϊόν, ένα εναλλακτικό. Λέτε ότι η επένδυση θα πάει σε διαρθρωτικά σχέδια κτλ. Ναι, εντάξει, μακροπρόθεσμο, ωραία, εφόσον λέτε καλά το προϊόν. Οπότε καταρχήν δεν υπάρχει αντίθεση εφόσον οι επενδύσεις και οι επανεπενδύσεις θα είναι πραγματικά στέρες και γερές, ναι, εφόσον βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άνοιγμα της αγοράς κτλ. Ναι, αν διατηρήσουμε τους μικρούς παραδοσιακούς ασφαλιστές και ναι, εφόσον οι μεγάλοι, θεσμικοί σχεδόν μεγάλοι ασφαλιστές, λειτουργήσουν παράλληλα για να επωφεληθούν από αυτό το προϊόν, αλλά οδηγήσει αυτό σε μείωση των εισφορών. Όμως υπάρχουν και πολλά αρνητικά που βλέπουμε εμείς αυτή την υπόθεση. Λέμε όχι αν το προϊόν αυτό θα συμμετέχει, αλλά αυτό θέλει και εικόνα, στην ε, Ένωση Κεφαλαιογορών. Όχι αν ε, κρίνεται και κρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι μόνο η αρχή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων που εποπτεύει. και πώς θα οριστεί το λειτουργικό πλαίσιο και όλα τα στοιχεία από την ΙΟΠΑ, δηλαδή θα κρίνει και θα κρίνεται. Τι θα γίνει τότε με τους μικρούς παραδοσιακούς ασφαλιστές. Έπειτα, μήπως είναι και για να καλυφθεί η μείωση της αγοραστικής δύναμης και το γεγονός ότι έχουν καταστεί τόσο ευάλωτα τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα. Θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές εξαιτία των ψηφιακών κτλ. Η απασχόληση ε, θα γίνει περισσότερο επισφαλής και θα υποφέρουν περισσότερο οι γυναίκες και οι πιο ευάλωτοι από αυτό. Οπότε, ε, πολύ ωραίες οι προθέσεις του συναδέρφου, εντάξει. Ε, ποιοι είναι αυτοί οι πιο ευάλωτοι, θα μπορέσουν αυτοί να πληρώσουν για να έχουν αυτή την παραπάνω σύνταξη, ή μήπω τελικά καταλήγει αυτό το συνταξιδοτικό προϊόν να είναι μια σύνταξη μόνο για τους πλούσιους και μόνο για αυτούς που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη σύνταξή τους Και τι θα γίνει με τα κοινωνικά συστήματα, μήπω πλήττονται επιπλέον και τα φορολογικά επίση, διότι κάποιες τροπολογίες προβλέπουν και φορολογικέ προτάσεις και λέμε επίσης όχι αν τελικά θέλουμε να βοηθήσουμε μόνο τους μεγάλους θεσμικούς ασφαλιστές, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς σε μερικές χώρες είναι περίπου μονοπόλιο. Και τελικά βρισκόμαστε σε αγορές με μονοπόλια, όπως το έχουμε δει σε μερικές περιπτώσεις, όταν αποφασίστηκε από χώρες και από κοινοβούλια να συμμετέχουν σε μια ομαδοποιημένη αγορά. Θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Θα υποβάλουμε πολλές τροπολογίες προς την κατεύθυνση που είπα. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι η Ευρώπη αυτή που πρέπει να πάει προς μη, η οποία τελικά είναι καθαρά εθνική και δεν θα έπρεπε να είναι ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πέκερ πάλι για να αντιδράσει στα όσα ακούσαμε. Παρακαλώ. Yes. Äh, okay. Sorry, Mr. Μια στιγμή, μια στιγμή. Συγγνώμη κύριε Δεμπάκερ. Κάποιος ζητά το λόγο. Η κυρία Πένια Γκονζάλες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, συγγνώμη που δεν ζήτησα το λόγο πριν. Ε, παρακολουθούσα μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις παρακαλώ για αυτό το πανευρωπαϊκό ατομικό σταξιδιωτικό προϊόν. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι εδώ δεν πρόκειται για έναν μηχανισμό κοινωνικής προστασίας, αλλά για μια επιπλέον ευκαιρία στην αγορά. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Κατά τη γνώμη μας, οι συντάξεις είναι και πρέπει να είναι θεμελιώδης δικαίωμα για να μπορεί κανείς να ζήσει ικανοποιητικά μετά την εργασία του. Είναι βασικό δικαίωμα για ολόκληρη την κοινωνία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το έργο μας πρέπει να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπών δημόσιων συντάξεων. Δεύτερον, λέμε ότι είναι ένα ιδιωτικό αυτό προϊόν, έτσι τι διαφάνεια θα υπάρχει στις επενδύσεις που θα γίνουν για αυτό το πανευρωπαϊκό προϊόν. Είναι απίστευτο. Ενώ η ζωή κρατάει περισσότερα χρόνια ακόμα, αντί να υπάρχουν χρήματα ε, στο δημόσιο και λέμε και ξαναλέμε ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις και τα λοιπά. Από την άλλη μεριά λέμε ότι δημόσιο χρήμα θα επενδυθεί σε ιδιωτικές συντάξεις. Γίνεται δηλαδή μια εμπορική συναλλαγή καθαρά. Εμείς θέλουμε ένα δημόσιο πανευρωπαϊκό ταμείο για τις συντάξεις που να προσφέρει αλληλεγγύη μεταξύ όλων των Ευρωπαίων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δηλαδή όχι εμπορικές συναλλαγές για τις μεγάλες οικονομικές οντότητες, αλλά να διασφαλίσουμε δημόσια σύνταξη για όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Υποβαθμίζουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, αυτό κάνουμε μέχρι τώρα και επειδή διαπιστώνουμε κάποια στιγμή ότι δεν λειτουργούν καλά, τις ιδιωτικοποιούμε. Ε, αυτό ακριβώς κάνουμε και με τις ασφάλειες τώρα. Δηλαδή, θα προωθήσουμε, θα προμοδοτήσουμε τις ιδιωτικές ε, συντάξεις. Γιατί, Γιατί υποβαθμίζουμε τις συντάξεις που προσφέρει το δημόσιο, λέμε ότι δεν είναι κανονοποιητικές, δεν λειτουργούν, δεν ε, εξυπηρετούν, οπότε φτιάχνουμε τις ιδιωτικές. Εμπόριο δηλαδή. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό το προϊόν. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε τώρα, κύριος Μπέκερ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε, ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω τώρα αυτά ε, τα ερωτήματα τα οποία ε, ε έλαβα αρχικά κυρία Γιουγκέριους εγώ ο ίδιος ε, είμαι άτομο ε, το οποίο υποστηρίζει την ε, αρχή της, του πρώτου πυλώνα. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι ξεκάθαρο. Ο δεύτερος πυλώνας επίσης ιδιαιτέρως επειδή ε, αναπτύχθηκε χάρη στις κάτω χώρες ε, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ε, ποιότητας ε, και έχουμε μια καλή μορφή διασφάλισης, συνταξιδιωτικής διασφάλισης. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι εδώ μιλάμε μονάχα για ένα επιπρόσθετο προϊόν, ένα προϊόν το οποίο μπορεί κάποιος να κάνει εθελοντικά. Και φυσικά θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε επιρροή στην πρώτη και, στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα των ε, κρατών ε, μελών. Ε, ήρεμα λοιπόν, ε, έχουμε, θα, είμαστε, θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι σε περίπτωση που υπάρξει ένα επιπρόσθετο προϊόν το οποίο ε, λύνει προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε αρκετές περιοχές των 28 κρατών μελών. Ε, σε περίπτωση ε, που δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, τότε με αυτό το προϊόν σε αυτές τις περιοχές μπορούμε να έχουμε μια πολύ θετική επίδραση. Θα ήθελα να επιβεβαίωσω λοιπόν άλλη μια φορά, είναι ξεκάθαρη γραμμή, ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας δεν θα ακουμπηθούν, αυτό το αναγνωρίζω, το ξεκαθαρίζω Όσον αφορά τώρα ε, την αξιολόγηση ε, της αποδοτικότητας του ΠΕΠ ύστερα από πέντε ε, χρόνια, αυτό το αποδέχομαι και θα περιμένω τις τροπολογίες. Ευχαριστώ για αυτήν την πρόταση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λίντάιερ ε, η οποία μίλησε ιδιαίτερως ε, για το ε, μακροπρόθεσμο κομμάτι του ΠΕΠ και ιδιαίτερως για το διασυνοριακό χαρακτήρα του ΠΕΠ, το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως είπαμε, η φορολογική εναρμόνιση και υπόθηκε ήδη ε, στο θέμα των φόρων ε, δεν μπορούμε να παρέμβουμε, ε, δεν υπάρχει αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Επιτροπή Απασχόλησης επίσης, όμως θέλουμε η διαπραγμάτευση να είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο έγινε και με άλλα προϊόντα. Από τον κύριο Σαμπού υπήρχαν θετικά σημάδια, το γεγονός ότι μπορούμε να το πάρουμε αυτό ως βάση, ωστόσο όσο αφορά τη διαφάνεια, την ασφάλεια, την ε, ε, δυνατότητα, τη δυνατότητα μεταφοράς ε, και, τον έλεγχο, και ο έλεγχος αυτός να βρίσκεται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην έχουμε νέες γραφειοκρατικές δομές σε εθνικά επίπεδα. Ε, συμφωνώ μαζί σας λοιπόν και χαίρομαι για αυτή σας την πρόταση. Για την κυρία τώρα από την ΚΟΥΕ, την κυρία Κούνεβα, το παρουσίασε τόσο τρομακτικά ότι δηλαδή σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης υπάρχουν συντάξεις οι οποίες δεν διασφαλίζουν ε, τα προστοζήν ε, εδώ ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούμε άμεσα να παρέμβουμε. Αυτό είναι ζήτημα των συνθήκων μεταξύ των ε, κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Θα επιθυμούσα να μπορούσαμε να το κάνουμε και να μπορέσουμε να ασκήσουμε περισσότερη πίεση. Ε, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται ήδη μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της Κομισιόν. Ε, θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ε, για το πρώτο και δεύτερο πυλώνα ε, ο κύριος Γκονζάλες ναι είναι ένα ε, προϊόν ε, της κεφαλαιογοράς όμως έχει μια κοινωνική διάσταση την οποία την τόνισα επανειλημμένως και έγκυται στους τομείς όπου δυστυχώς δεν υπάρχουν κοινωνικά συστήματα συντοξιοδότησης έτσι λοιπόν αυτό το προϊόν της αγοράς θα είναι μια πολύ καλή υποστήριξη για εκατομμύρια ανθρώπους ανθρώπους ανά την Ευρώπη. Ε, για την ε, κυρία από το ENF ε, τόνισε ότι ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας είναι ένα σημαντικός ε, παράγοντας ε, και θα πρέπει να διασφαλίζεται από, το όσο, όσο το δυνατόν περισσότερους παρόχους. Ακόμα και μικρότεροι ασφαλιστές θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ναι, θεωρώ ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Πολλούς από τους παράγοντες δεν τους βλέπω ως πρόβλημα, αλλά παρακαλώ καταγράψτε τις σκέψεις σας και θα τις συζητήσουμε συζητήσουμε. Όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των συντάξεων, δεν συζητάμε κάτι τέτοιο τα κράτη-μέλη μόνα τους αναπτύσσουν τα συνταξιδοτικά τους προγράμματα και από αυτήν την πρωτοβουλία της Κομισιόν, την οποία διαπραγματευόμαστε εδώ πέρα, δεν μιλάμε για, ε, για ιδιωτικοποίηση των ε, συνταξιοδοτικών συστημάτων. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις ε, προτάσεις σας, χαίρομαι για την συνεργασία που θα έχουμε. Υπάρχουν δύ... άλλες δύο-τρεις συναντήσεις των σχεδόν, όπου θα τα συζητήσουμε αυτά αυτά παρόλο που είναι σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έχει έρθει η κυρία ε, Μπάλιγκε από την Κομισιόν. Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Κομισιόν για την υποστήριξη του εισηγητή καθώς και για τους ευρωβουλευτές για τα καλά τους λόγια όσους παρενέβησαν υπέρ αυτής της πρότασης. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε σχέση με τη φύση αυτής της πρωτοβουλίας. Όπως είπε και σωστά ο κ. Μπέκερ, ο στόχος δεν είναι να παρέμβουμε στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι συντάξεις στα κράτη-μέλη αυτή δεν σχετίζεται με τον πρώτο πυλώνα και τις κρατικές συντάξεις, ούτε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβατικές ε, οι συμβατικές, ε, συμβατικά μάλλον συνταξιδοτικά ταμεία, αλλά ε, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ε, Μάλλον, στόχος είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ε, εθελοντικό ε, πρόγραμμα. Δεν υπάρχει υποχρέωση ε, για κανέναν πάροχο και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ε, για κανέναν πολίτη να πάρει το ΠΕΠ. Εμείς σκεφτόμαστε εκείνους τους πολίτες που βρίσκονται στα κράτη-μέλη όπου το επίπεδο παροχής ε, των συντάξεων ε, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Σκεφτόμαστε πώς θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του και χάσματος των συντάξεων, να καταθέσουμε δηλαδή μια πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του, της διαφοράς μεταξύ των φύλων. Επίσης σκεφτόμαστε τις περιπτώσεις ε, των κινούμενων πολιτών στην Ευρώπη γιατί το ΠΕΠ θα είναι πραγματικά πανευρωπαϊκής φύσης και θα είναι δυνατόν ε, για τους πολίτες ε, που μένουν στην Ένωση, να οπουδήποτε στην Ένωση, να συμβάλλουν στο συνταξιδοτικό αυτό μέσο. Θα θέλαμε όλοι οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα απλό, διαφανές και αποτελεσματικό προσωπικό συνταξιδοτικό προϊόν. Να μπορούν να αναπτύξουν τις οικονομίες τους. για τα γεράματά τους και κυρίως σκεφτήκαμε αυτούς που ε, έχουν ε, σχετικά χαμηλά εισοδήματα. Εμεί ε, θα περιμένουμε τις πρότασεις σα για βελτιώσει. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τις ομάδες ε, στην ΕΚΟΝ, στην ΕΜΚΟ και στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για να συμβάλλουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε πως οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το προϊόν σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση αυτή είναι η προθεσμία δηλαδή για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 7 Μαΐου τις 12 το μεσημέρι, η έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης 28 Ιουνίου, στην ΕΚΟΝ 11 Ιουλίου και θα περάσει από την Ολομέλεια, δεν ξέρουμε πότε, θα επιβεβαιωθεί αργότερα. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας και περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019. Εντολή για τον τριμερή και ανταλλαγή απόψεων. Ως ε, εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης για τον Προϋπολογισμό με χαρά βλέπω ότι ο αγώνας κατά της νεανικής ε, ανεργίας έχει αναγραφεί ως πρώτη πρόκληση και προτεραιότητα για την Ένωση, καθώς και στις κατευθύνσεις γραμμές του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 19. Επίσης θα ήθελα να ε, θερμά, θερμά το ενέμφαση που δίνεται στην ανάγκη να αναπτυχθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες και να υπάρχει μηδένα αναγνώριση των δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου. Αναμένουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες ακόμα για, ε, και προτάσεις για να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων στο σχέδιο της γνωμοδότησής μου λέω γενικότερα πως ο προπολογισμό του 19 θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των του, του στόχου του 2020 καθώς και την επιτυχή εφαρμογή των νεότευτου πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και της μης ανεργίας, αλλά και ε, την εξέβρεση λύσεων και την για, την για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για το, 1900, ε, το 2019 ε, δεν προβλέπονται περικοπές από ό,τι φαίνεται ούτε στο PDP. Ε, γιατί κάτι τέτοιο θα υπέσκαπτε τις πολιτικές μας δεσμεύσεις και πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. Από αυτό κρέμεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ζητώ ως εισηγήτρια να διατηρήσουμε αυτές τις γραμμές. Να θυμίσω και το σημαντικό έργο των διαφόρων οργανισμών στο δικό μας τομέα, Eurofund, OSHA, SEDEFOP, και τα περασμένα χρόνια χρειάστηκε σημαντική προσπάθεια από πλευράς τους παράγραφο 20 του ψηφίσματός μας να θυμίσω ότι ζητάμε να μην υπάρξει άλλη περικοπή στους πόρους για το 19. Τέλος, ορισμένα ε, σημεία θα έρθουν για αξιολόγηση από πλευράς ε, της Επιτροπής μας και νομίζω πως είναι αυτό ένα καλό μέσο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για καινούριε και γενοτόμε ιδέε. Α πούμε, η πρόταση για την εγγύηση για τα παιδιά είναι ένα παράδειγμα που έρχεται τώρα εύκολα στο μυαλό μου και ζητώ το Κοινοβούλιο να, δίνεται, να, να λαμβάνει τακτική και λεπτομερή ενημέρωση για τα διάφορα στάδια της εφαρμογής των πιλωτικών ή των προπαρασκευαστικών δράσεων από την Κομισιόν. Και βεβαίως η Κομισιόν οφείλει να σέβεται το περιεχόμενο που πως το έχει εγκρίνει η Δημοσιονομική Αρχή. Και θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα σχόλιο για την φάση εξολόγησης, όπου είναι σημαντικό οι προτάσεις να δίνονται στις σωστές Γενικέ διευθύνσει τη Κομισιόν είχαμε κάποιε κακέ εμπειρίε τα τελευταία χρόνια, ότι δηλαδή οι προτάσει βαθμολογούνται με τη βάση μόνο της, της, του τους. Γι' αυτό και εγώ ζητώ λεπτομερεί προτάσει. Δηλαδή κάποιες γενικές γραμμές δεν αρκούν και σε περίπτωση που όπως πέρυσι κάποιοι συνάδελφοι αντιμετώπισαν προβλήματα και αναγκάστηκαν να περάσουν από διάφορες γενικές διευθύνσεις και διαπιστώσαμε πως τα τελικά κάποια πιλωτικά προγράμματα και κάποιες προπαρασκευαστικές δράσεις δεν είχαν αξιολογηθεί σωστά ε, και ζητήσαμε να επαναξιολογηθούν υπό το φως αυτών των σφαλμάτων που είχαν γίνει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βιώτη που είναι ο Γενικός Συγητής για το προπολογισμό του 2019. Αν έχετε κι εσείς κάποια σχόλια να μας κάνετε από τώρα σε αυτό το πρώιμο στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή που με κάλεσε, την Επιτροπή σας που με κάλεσε σε αυτή τη συζήτηση και για τη σημαντική συμβολή που έχετε ήδη κάνει στην περίπλοκη μου αυτή ε, δουλειά για φέτος. Συμφωνώ με απόλυτα με τα όσα προτείνει η Επιτροπή σας. Εφόσον το ψηφίσετε θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε και τις κατευθύνσεις γραμμές για, τον επόμενο, για προπολογισμό του επόμενου χρόνου που το ψηφίσαμε το Μάρτιο και θα έχετε εκτιμήσει το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε το θέμα το κοινωνικό αλλά και το θέμα της απασχόλησης το τονίσαμε ιδιαίτερα στις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Τώρα, δύο θεματολογικές παρατηρήσεις και μετά επί της ουσίας. Για τη μέθοδο γνωρίζετε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι πολύ άκαμπτος. Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν επιτρέπει να κάνουμε περιοέτες, ούτε να είμαστε φάνταστοι στο να εφευρίσκουμε καινούργια πράγματα. Μας υποχρεώνει να εργαζόμαστε σε γραμμές που ήδη υπάρχουν. Ωστόσο, ζητώνται και εμείς κάποιες φορές ε, τα στηρίζουμε όλα αυτά ε, και ζητώνται νέες πρωτοβουλίες από πλευράς των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Σε άλλες επιτροπές μιλήσαμε για άλλα project, για την άμυνα κτλ. Αλλά πιστεύω πως είναι ένα επιχείρημα το οποίο αφορά πολύ ε, στενά τη δική σας επιτροπή, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ε, και το στηρίζουμε και το προωθούμε. Είμαστε όμως ε, πεπισμένοι πως χρειάζονται νέοι πόροι, ότι δεν μπορεί διαρκώς να έχουμε έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό όπου περικόπτονται οι, οι πόροι και απλώς γίνονται μεταφορές προς νέες γραμμές. Αυτό είναι εις βάρος της ε, σοβαρότητας του προϋπολογισμού και αποθαρρύνονται οι πολίτες που είχαν ε, προσδοκίες για τον προϋπολογισμό. New fresh money χρειαζόμαστε. Και προχωρώ πολύ γρήγορα για ορισμένους από τους προβληματισμούς και τις παρατηρήσεις της, της Προέδρου. Διότι συμφωνώ απόλυτα πέρυσι, Όντω χάρη στην εργασία του προκάτοχού μου, του εισηγητή μου Ρεσάν, έγινε σημαντική δουλειά όσον αφορά την εγγύηση για τους νέους και μπορέσαμε να καταφέρουμε σε δύσκολες διαπραγματεύσεις ένα σημαντικό, μια σημαντική αύξηση για φέτος. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε σε αυτήν την ε, ωραία πορεία και να αποφύγουμε να υπάρξουν περικοπές στα διάφορα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, την πρωτοβουλία για τους νέους, τα χρήματα για την αντιμετώπιση της ε, παγκοσμιοποίησης, ε, ο αγώνας κατά της φτώχειας κτλ. Να προσπαθήσουμε δηλαδή ακόμα και να ανακτήσουμε κάποια χρήματα και θα κάνω και μια παρατήρηση πολιτικής χαρακτήρας αφού είμαστε στο Κοινοβούλιο, πολιτική κάνουμε εδώ. Πιστεύω πως η εικόνα που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη, τα τελευταία δέκα χρόνια, είναι μια εικόνα μιας ε, γρινιάρας και τσιγκούνα Ευρώπης εικόνα έχει δώσει. Ζητά συνέχεια ε, λιτότητα, αυστηρότητα, περιορισμό, σφίξε τα και πρέπει τώρα να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα γιατί οι λαϊκισμοί καταπολεμώνται με την καλή πολιτική και όχι με άλλους λαϊκισμούς ή με ευρωπαϊστικές ιδέες που είναι μόνο βιτρίνα. Λοιπόν, θέλετε στο σχέδιο γνωμοδότησής σας το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται διαρκώς από την Κομισιόν σε σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Φυσικά αυτό θα το μεταφέρω, θα το διαβιβάσω στον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο που θα έρθω σε επαφή μαζί του την επόμενη φορά. Μάλιστα δικαίως αναφέρεστε και σε την προσαρμογή των πληρωμών για το 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που σήμερα δεν λειτουργεί, δεν, μάλλον δεν απορροφά πλήρως του πόρου, αλλά θα φτάσουν διάφορα project που θα πρέπει να εξοφληθούν και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κρίση πληρωμών όπως είχαμε το 2014. Για τους οργανισμούς συμφωνώ απολύτως για όλους τους οργανισμούς ζητάμε νέες δεσμεύσεις, νέες, ε, νέες, ε, νέα καθήκοντα, αλλά απ' την άλλη μιλάμε όλο για περιορισμούς και περικοπές του προϋπολογισμού. Ε, πρέπει να μπορούμε να έχουμε νέους ε, πόρους, όπως και για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους διάφορους οργανισμούς, εφόσον τους ζητάμε συνέχεια και τους αναθέτουμε νέα καθήκοντα. Τώρα, Τέλος, για την προπαρασκευαστική συγγνώμη δράσεις. Ε, θέλω να είμαι σαφής. Ε, έχω μεγάλο σεβασμό στη δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπάλληλοι τη. Ε, όσον αφορά την αξιολόγηση των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων, PP και PD κάνει ε, πολλή δουλειά η Κομισιόν, αλλά εμείς ε, πρέπει να μπορούμε να εκφράσουμε τις πολιτικές μας επεπιθήσεις. Ε, το πέρυσι έγινε και αν υπάρξουν πιλωτικές, πιλωτικά προγράμματα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητα γιατί ο καλό των συμπολιτών μας και υπέρ των κοινωνικών πολιτικών πρέπει να γίνουν, εγώ θα τη εντάξω στο πακέτο. στις γραμμές για τις δράσεις, ε, τις έκτακτες δράσεις μεγάλης σημασίας. Αυτά λοιπόν και περιμένω τις περαιτέρω σας ε, παρατηρήσεις ε, και δεσμεύομαι να δουλέψουμε πλάι-πλάι σε αγαστή συνεργασία μέχρι την τελευταία στιγμή και την τελευταία ημέρα της συνδιαλλαγής. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη και για τα όσα είπατε μέχρι τώρα. Η κυρία Γιονγκέριος τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το εξαιρετικό σας σχέδιο που υποβάλλατε σήμερα και για την παρουσίαση που μας κάνατε της κατάστασης πρόοδου στην δική σας Επιτροπή. Μας βοηθά πολύ στην συζήτηση. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους είναι σημαντικός για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του 2020. Όμως εδώ πρέπει να θυμόμαστε πως και η δημοσιονομική ευελιξία χρειάζεται ώστε να στηριχθούν κοινωνικές επενδύσεις και κοινωνικά δικαιώματα. Χρειάζεται ο προπολογισμό, αλλά χρειάζεται και η δημοσιονομική ευελιξία. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ε, και όταν λέω εμείς συμφωνούμε, εν, το λέω γιατί χρησιμοποιώ τα σημειώσει του κυρίου Πριέτο που είναι ο σκιώδης μας. δυστυχώ δεν μπορούσε να είναι εδώ παρόν γιατί είναι ζεροπλάνο κάπου μεταξύ Ισπανίας και Βρυξελών. Έχουμε λοιπόν νεότητα, απασχόληση, ισότητα, καταπολέμηση αποκλεισμού και φτώχε. Αυτά, αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις και μπορεί να τελειώσει αυτή η εντολή ενώ δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτοί. Ο Σέρζιο θα εξετάσει την ε, δυνατότητα για τις βασικές μας δεσμεύσεις πρέπει να δουλέψει η Ευρώπη για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της, σε, σε ολόκληρη την επικράτεια και τα παιδιά είναι αυτά που υποφέρουν περισσότερο, είναι τα πιο ευάλωτα από τέτοιε καταστάσεις. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τελειώσουμε αυτή την εντολή χωρίς ένα σαφές μήνυμα και δέσμευση πω το ευρωπαϊκό project λειτουργεί και για Κίνα και να τους προστατεύσουμε και να τους προσφέρουμε καλύτερες ευκαιρίες στην ζωή. Γι' αυτό και ε, υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χάρτη για τα παιδιά να συνταχθεί αυτός όσο γίνεται πιο σύντομα και μάλιστα έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά πολύ. Η βιώσιμη δε ανάπτυξη δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς να υπάρχει μια ε, ε, ευημερία η οποία κατανέμεται σε όλους τους πολίτες και φτάνει σε όλους τους πολίτες. Ε, θέλουμε να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2020-2030 και οι βιώσιμοι στόχοι, αλλά ε, θα πρέπει να προωθήσουμε και προς τα πάνω την κοινωνική σύγκληση. Αυτό μπορεί μόνο να επιτευχθεί με ισορροπημένους ισορροπημένες πολιτικές ανακατανομής του οι ανισότητες ε, δεν μπορούν ε, ως διαθαύματος να διορθωθούν, να ε, <coughs> καλυφθούν. Γι' αυτό και θα πρέπει να φτιάξουμε και έναν δίκτυο κοινωνικής πρόοδου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο για την αξιολόγηση της επιτυχίας της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην επίτευξη καλύτερων κοινωνικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους οργανισμούς γνωρίζουμε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Απασχόληση και αυτή θα απαιτήσει και άλλα χρήματα. Αλλά ανησυχούμε πολύ για τη δυνατότητα τη πιθανότητα μάλλον περικοπής των προϋπολογισμών άλλων οργανισμών, γιατί αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα της εργασίας που κάνουν αυτοί οι άλλοι οργανισμοί και να ε, απειλήσει τη λειτουργία τους μάλιστα. Ζητούμε λοιπόν από την Κομισιόν να εξετάσει προσεκτικά τον προϋπολογισμό και να ε, γίνουν ε, προσπάθειες ε, συνδυασμένες με φρέσκα χρήματα και αυτή η επιλογή είναι η προτιμότερη από οποιαδήποτε περικοπή σε οποιονδήποτε προϋπολογισμό οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Τώρα, Πρέπει να προσέξουμε και τις γραμμές εκείνες που είναι αφιερωμένες στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Γιατί έχουν διατυπωθεί ανησυχίες από τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά την ανεπάρκεια των κονδυλίων που αφιερώνονται στο κοινωνικό διάλογο και στα project των κοινωνικών εταίρων και δεν μπορούμε από τη μια πλευρά να δηλώνουμε ότι είμαστε προσιλωμένοι στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, να ζητάμε από τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετέχουν περισσότερο στο εξάμεινο ενώ στην εφαρμογή των πολιτικών και στην εφαρμογή μάλλον των πολιτικών, ενώ ταυτόχρονα δεν εξασφαλίζουμε ε, δημοσιονομικά τη λειτουργία τους. Και σε αυτές τις γραμμές θα προετοιμάσουμε και τις προτάσεις μας ε, για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. ευχαριστώ ε, πολύ. Ε, του χρόνου, το 2019 λοιπόν, θα είναι η χρονιά ε, που η Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή η πολιτική αλλαγή θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ε, προβλήματα προσαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερω εφόσον η Μεγάλη Βρετανία συνεισφέρει έντονα ε, στον προϋπολογισμό της Ένωση. Ε, μιλάμε για προστιθέμενη αξία. Όμω, πολύ συχνά υπάρχει επιθυμία για πιο σοβαρή διαχείριση των χρημάτων. Για παράδειγμα θα ήθελα να σας μιλήσω την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων πέρσι, το ε, το ελεγκτικό συνέδριο ε, δήλωσε ότι υπάρχουν ε, προβλήματα με αυτό. Ε, μιλάμε για χρήματα, για χρήματα των πολιτών της ε, Ένωσης. Ε, κάθε πρόγραμμα, όσο ωραίο και αν είναι το όνομα, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να του ρίχνουμε χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν πιο συνειδητά να διαχειριζόμαστε τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών και ειδικά όταν μιλάμε για προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με όλα αυτά. Τα κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένα προβλήματα και σε μια εποχή που έχουμε ε, χαμηλότερη οικονομική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή, ε, στην Ευρωζώνη και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένες ε, λύσεις και όχι απλά έτσι να ρίχνουμε χρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα της επικουρικότητας είναι ξεκάθαρο στις συνθήκες και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το προσέχουμε περισσότερο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τα βοηθήσουμε ώστε να μην χώνουν τα, χρήματά τους σε κοινωνικά προγράμματα, αλλά σε προγράμματα τα οποία δημιουργούν ε, ανάπτυξη, επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων, ε, εργασίας, ε, να βοηθήσουμε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, διότι ε, ε, θα πρέπει όλα αυτά λοιπόν να εξεταστούν διότι ε, δεν γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματικά είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2019 θα είναι η χρονιά που η, Μεγάλη Βρετανία θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι μια καλή στιγμή να αναλογιστούμε και εσείς κυρία εισηγήτρια για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτή τη σοβαρή κρίση διότι μιλάμε για ε, ε, περικοπές ε, ή είναι άλλα τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Θα Προσπαθούμε λοιπόν με τις τροπολογίες μας να δώσουμε τα κίνητρα για κάτι τέτοιο και θα χαρώ να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν από την Άλντε. κανένας από την Άλντε που ζητάει το λόγο. Η κυρία Λαμπέρτ, λοιπόν, ευχαριστώ ε, πολύ ε, και συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε η κυρία Τρεπέσιους η Μεγάλη Βρετανία ε, φεύγει ε, μπορεί ε, να γίνει μια αξιολόγηση στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε την διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο κόσμος συνειδητοποιεί το τι θα χάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ακρόαση ε, στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ε, δηλώνει πως θα κάνει αντικαταστάσεις, όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο και υπήρχαν προσπάθειες έντονης προστιθέμενης αξίας, όχι μονάχα με ό,τι συνέβαινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και με τη δυνατότητα να μαθαίνουμε από άλλους. Βλέποντας λοιπόν την προστιθέμενη αξία δεν είναι μονάχα ε, θέμα ε, που αφορά ε, τις λεπτομέρειες του προγράμματος αλλά γενικότερα τη μεθοδολογία αυτών των προγραμμάτων, τις εταιρικέ σχέσεις, το ότι φέρνουν κόσμο να συνεργαστεί και το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί πιο ευρύτερα. Τώρα όσον αφορά τον ε, προϋπολογισμό για του χρόνου και όχι το ε, πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα θέλουμε να πούμε ότι συμφωνούμε γενικά με τον εισηγητή, με την εισηγητρία, ότι πιστεύουμε μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2020 για την απασχολησιμότητα, την εφαρμογή του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων όσον αφορά τώρα τα ποσά τα οποία αναφέρθηκαν ε, και τα ταμεία τα οποία αναφέρθηκαν θα θέλουμε να τα ε, κρατήσουμε. Ε, αυτή είναι, όπως είναι η γνώμη της συγγήτριας. Υπάρχουν ακόμα οι ανάγκες και συνολικά η θέση μας είναι ότι υποστηρίζουμε να συνεχιστεί η υποστήριξη στο κοινωνικό ταμείο και ιδιαίτερως όσον αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ε, όσον αφορά την αρχή εργασίας ε, και εκεί θέλουμε να εξετάσουμε πώς μπορεί να ταιριάξει όλο αυτό. Εξετάζουμε, το εξετάσαμε αυτό όταν κάναμε ε, το έργο για το σώμα των εθελοντών ε, και εκεί έχουμε διάφορα ε, προγράμματα τα οποία είναι πολύ ε, αποτελεσματικά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από εκεί σε άλλους τομείς, σε γενικές γραμμές λοιπόν ο προϋπολογισμός μας αφορά ιδιαίτερος, ιδιαίτερος όσον αφορά την υποστήριξη και ε, συμφωνούμε με τα όσα υπόθηκαν από, το, ε, ε, από τους συλλιστές όσον αφορά την αποσχολησιμότητα, όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, έγιναν κάποια σχόλια, όμως για κάποια διαλύματα σε διάφορα πιλωτικά προγράμματα τα οποία προτάθηκαν, το υποστηρίζουμε και εμείς αυτό και υπάρχουν, προωθούμε κάποιες ιδέες ε, από αυτήν την Επιτροπή αλλά και από το Κοινοβούλιο ε, που προτείνονται εδώ και καιρό. Αυτή είναι η γενικότερη προσέγγιση όσον αφορά την ε, γνωμοδότηση. Βέβαια θα υπάρξουν κάποιες τροπολογίες, όμως θεωρούμε ότι η γενική κατεύθυνση της συγγήτριας μας βρίσκει σύμφωνος. Ευχαριστώ πολύ. Από το FTD, η FTD δεν είναι κανένας. ο κύριος Ντομινίκ Ματών από το ε, EMF. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν εκπλήσει κανέναν φαντάζομαι, αλλά δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας. Γιατί όσο περνούν τα χρόνια, ο προπολογισμό του 2019 είναι ακριβώς το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνει τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο, το 2015, το 2016, το 2017 και για το 2019 και για τους στόχους 2020. Αυξάνει η ανεργία, οι νέοι δεν έχουν δουλειές, οι μικρές επιχειρήσεις στραγγαλίζονται, δεν ε, ε, μειώνεται η ανεργία, οι εργαζόμενοι δεν καταφέρνουν ε, με τους μισθούς τους να ζουν ε, αξιοπρεπώς, οι άνθρωποι όλο και περισσότερο ζουν μέσα στη φτώχεια και αυτά κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια. Και αντί να αντιμετωπίζουμε τις αιτίε που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, προσπαθούμε τις συνέπειες να τις διορθώσουμε κάπως με εκατομμύρια που κάθε χρόνο βάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα τα οποία όμως βγαίνουν από τις τσέπες των συμπολιτών μας. Μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της παγκοσμιοποίηση, Εντάξει, το ψηφίζουμε γιατί είναι ένα τρόπο, εμεί οι Γάλλοι τουλάχιστον αυτό θέλουμε, να μπορούμε να ανακτούμε τα χρήματα, αλλά το σύστημα είναι ανόητο. Πληρώνουμε για θέσει απασχόληση που εμεί ήδη καταστρέφουμε. Έπειτα υπάρχει κοινωνική καινοτομία. Το είπαμε και αυτό είναι γελίο. Το Ταμείο ε, για τη βοήθεια απέναντι στους πιο φτωχούς. Και αυτό είναι γελίο. Οι πρωτοβουλίες για τους νέους. Το ίδιο το λεκτικό συνέδριο λέει ότι είναι μια καταστροφή και εσείς θέλετε όλο και περισσότερα χρήματα να βάλετε μέσα σε αυτό το ταμείο. Οι διαπιστώσεις είναι ίδιες κάθε χρόνο και τίποτα δεν αλλάζει. Θέλω να πω και στου εκπροσώπου τη Επιτροπή δεν ήρθε η στιγμή να θέσετε τα σωστά ερωτήματα. Εμείς το λέμε εδώ και χρόνια. Δεν είσαστε εκπρόσωπος της Επιτροπής, όχι. Α. Και έπειτα, πολύ πολιτικά θέλω να σας τα αναφέρω όλα αυτά. Μ' άρεσε αυτό που είπατε. Α, είσαστε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Α, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θέλετε να αγωνιστείτε κατά των λεκισμών. Αυτή είναι η προτεραιότητά σας. Μα κύριε, αντιλαμβάνεστε ότι ο λαϊκισμός, όπως το ονομάζετε, είναι η δημοκρατική έκφραση των λαών. Και αυτό θα έπρεπε να ήταν η προτεραιότητά σας. Αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι θέλοντας να καταπολεμήσετε το λαϊκισμό, όπως λέτε, τον τροφοδοτείτε και η πολιτική σας που έχει καταστροφικά αποτελέσματα και που προτείνετε την ίδια και την ίδια κάθε φορά είναι και η αιτία της αντίδρασης αυτής των λαών. Ωραία, συνεχίστε κύριε. Στο ίδιο μοτίβο και θα δείτε τι θα γίνει με τον λαϊκισμό. Κάποια στιγμή θα σας αντικαταστήσει. Πολύ απλά. Και μάλιστα πολύ γρήγορα θα συμβεί αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα να αντιδράσει και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Η κυρία Φελάη, τμήματάρχη, σωστά. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτό το στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα τη δράση στην πρόταση. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για το σχέδιο που έχετε ετοιμάσει. Στηρίζουμε βεβαίως τόσα λέτε. Συμφωνούμε ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, συμφωνούμε ότι μένει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2020 σε διάφορους τομείς την ε, κοινωνική ένταξη, τη μείωση της ανεργίας των νέων κυρίως κλπ. Ελπίζουμε ο προπολογισμό 2019 να βοηθήσει να ενισχυθεί ο κοινωνικός ε, πυλώνας. Χαιρόμαστε για τη στήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτό και θα φροντίσουμε μαζί ο επόμενος προπολογισμό να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Να πω δύο λόγια για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Έχουμε μιλήσει και αυτά στην Επιτροπή σας πρόσφατα. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Αν νομίζετε ότι θέλετε πιο τακτικά ενημέρωση για αυτά τα δύο. Το έργο της Επιτροπής τώρα που κάνει αξιολόγηση είναι μια προσεκτική αξιολόγηση βάσει κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν συμφωνηθεί. Και οι κατηγορίες αντιστοιχούν σε πολύ σαφείς καταστάσεις. Μπορεί μερικές φορές να υπάρχουν επικαλύψεις. Όπως είπε και ο εισηγητής από την Επιτροπή προπολογισμών μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί εμείς κάνουμε την αξιολόγησή μας περισσότερο νομικά και τεχνικά, ενώ εσεί έχετε μια περισσότερο πολιτική οπτική γωνία. Αλλά σίγουρα πρέπει να καταλήξουμε στην ίδια αξιολόγηση. Θα την κάνουμε λοιπόν από τη δικιά μας την πλευρά και μετά θα τη συζητήσουμε φυσικά. Κάποιες προτάσεις μερικές φορές κυκλοφορούν μεταξύ διαφόρων γενικών διευθύνσεων γιατί ε, υπάρχει επικάλυψη μεταξύ διαφορετικών πολιτικών. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε ποια θα είναι η πιο κατάλληλη γενική διεύθυνση για να ελοπίσει τις προτάσεις σας. Πάντως πάντα στο τέλος βρίσκουμε λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βιώτη που θα πρέπει να ξαναπώ ότι είναι ο Γενικός Εισηγητής του Κοινοβουλίου για το 2019. Έτσι, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισηγητής. Λοιπόν, παρακαλώ, ποιες είναι οι αντιδράσεις σας όσο ακούσατε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι και ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μεγάλη χαρά μου έδωσε που άκουσα τις παρεμβάσεις ακόμα και τις πιο επικριτικές γιατί διαβλέπω τη βούληση να δουλέψουμε θετικά επικοδομητικά προτείνοντας από τώρα συμβολή με τροπολογίες, ε, συμβολή με ε, αναλύσεις και προβληματισμό. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι μεγάλη η ευθύνη και ρόλος που έχω αναλάβει να προσπαθήσω να αντιπροσωπεύσω ολόκληρο το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή όλους τους Ευρωπαίους ε, πολίτες και όλες τις ευαισθησίες που υπάρχουν. υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία είμαστε σε απόλυτη συμφωνία. Απλά θα ήθελα εγώ τώρα να μιλήσω για κάποια στοιχεία διαφορετικά ε, εκεί όπου διαφέρουμε, κυρίως δηλαδή αυτά που μας είπε ο συνάδελφος ε, Τρεπέζιος, ας πούμε για τη συνέπειες του Brexit για το 2019, Δεν θα υπάρξουν άμεσες ε, επιπτώσεις για το 2019. Η για το νέο πλαίσιο, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουμε πρόβλημα και θα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την Επιτροπή του Προϋπολογισμού και εν γέννη ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ φοβήθηκα πολύ ότι θα είχαμε ήδη πολύ βαριές συνέπειες στον προϋπολογισμό μας λόγω του Brexit. Αλλά ευτυχώς δεν είναι έτσι. Συμφωνώ με την ιδέα ότι και καταλαβαίνω το σκεπτικισμό σε σχέση με κάποια προγράμματα ε, όπως το το λογαριασμό για τους άπορους, ε, το Ταμείο για τους άπορους Υπάρχει το Ταμείο για τους Άπορους, ε, ε, υπάρχει το Ταμείο Προσαρμογής στην ε, παγκοσμιοποίηση και γενικά είχε θετικές, θετικά αποτελέσματα. Και το λέω και ως ε, εκπρόσωπος μια χώρας που χρειάστηκε να ζητήσει την ε, παρέμβαση του Ταμείου της ε, Παγκοσμιοποίησης λόγω πολλών μετακαταστάσεων. Και στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν θετικά τα αποτελέσματα. Οι υποθέσεις που εγώ παρακολούθησα στην Ιταλία, Whirlpool και άλλες υποθέσεις, ήταν πολύ θετικό και σε εξελίξεις και η χρήση ε, του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση. Όσον αφορά την εγγύηση για τους νέους, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, Καταλαβαίνω πως γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα και είναι αλήθεια πως το ελεκτικό συνέδριο τόνισε κάποιες ε, ε, κάποια προβληματάκια που υπήρξαν. Όμως αντιμετωπίστηκαν από την Επιτροπή Κοντ που σημείο προς σημείο απάντησε στα όσα είπε το ελληνικό συνέδριο. Να σας πω κάτι από τα παρασκήνια της φάσης ε, της συνδιαλλαγής της περασμένης χρονιάς δεν ξέρω αν είχατε τρόπο να συμμετέχετε στην ε, συνδιαλλαγή. Είναι αυτή η τελετουργία όπου βρίσκεται το Συμβούλιο σε μια αίθουσα, το Κοινοβούλιο σε μια άλλη και βέβαια εμείς ε, θα βασιστούμε πολύ, όπως ξέρετε και με το συνάρφο μου Ρεζάν πέρσι, ήταν υπέρ μια σημαντική αύξηση για την εγγύηση για τους νέους. Και εκεί το Συμβούλιο ήρθε τότε και μας είπε σε μια φάση ότι ε, κοιτάξτε έχουμε νέα από αυτές τις κυβερνήσεις μας είπε τις τάδε χώρες, ε, όπου δεν λειτουργεί καθόλου. Δεν υπάρχει καμιά παρόφηση. Ε, καθώς η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται και από μέλη α, και από αυτές τις χώρες που ανέφερε, εμείς επαληθεύσαμε με το αρμόδια Υπουργεία της εκάστοτε χώρας και μας είπαν ότι ναι, ήταν αληθινά τα στοιχεία. Διακόπτη πρόεδρος, χωρίς μικρόφωνο. Α, όχι πρόεδρο, συγγνώμη. Πόσο υψηλή είναι ε, το ποσοστό ανεργίας ε, στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Συγγνώμη, ε, θα ήθελα να σας πω ότι ε, τα χρήματα ε, μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν πολύ καλά από τις κυβερνήσεις, όμως παρόλα αυτά στη χώρα σας, στην Ισπανία, την Ελλάδα, άλλαξε με κάποιο τρόπο η ανεργία των νέων. Όχι, τα ποσοστά παραμένουν πάρα πολύ υψηλά και δεν θεωρώ ότι μπορούμε να το λυπηλήσουμε δίνοντας περισσότερα χρήματα, αλλά αρχικά θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ώστε να δημιουργηθούν νέες, νέα ποσοστά ανεργίας. Όταν στην Ελλάδα έχουμε ποσοστά ανεργίας, μεταξύ των νέων κα άνω των 60% ε, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Έχουμε δηλαδή μια διαφορετική οπτική γωνία σε όλο αυτό. Όχι, όχι. Και σας ευχαριστώ γιατί μου επιτρέπετε έτσι να εμβαθύνω περισσότερο ακόμη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, Ισπανία, Ιταλία, η νεανική ενεργεία βρίσκεται, ε, σιγά σιγά βέβαια, αλλά βελτιώνεται η κατάσταση. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ε, ότι η ανεργία είναι ανική, αλλά και η μη κοινωνική γενικότερα ε, λύνεται με παρεμβάσεις δημόσιες υπέρ των ε, ε, αναζητούντων εργασία αλλά κυρίως με δεσμεύσεις και επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση. Γι' αυτό το λόγο και αναφέρθηκα αρχικά και βέβαια δεν είσαστε εσείς αρμόδια επιτροπή, αλλά έλεγα ότι εγώ είμαι υπέρ ε, της διατήρησης των δεσμεύσεων ε, για τα μεγάλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το COSME, το Horizon 2020, το CEF, που δίνουν πραγματική βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνουν ε, βοήθεια στις, στα ερευνητικά ιδρύματα, στις επιχειρήσεις μας εν γέννη. Ε, να δουλέψουμε δηλαδή σε διαφορετικά μέτωπα. Ε, ε, να έχουμε δηλαδή ένα σύστημα πρόνοιας που να εγγυάται την προσαρμογή των νέων και στην τρόπο εργασίας που αλλάζει. Δηλαδή να έχουμε μια βιομηχανία που ανανεώνεται αλλά ταυτόχρονα μέσα τα οποία να είναι για την απασχόληση που να είναι εξυγχρονισμένα, να μην είναι τα μέσα που έχουν μείνει στην δεκαετία του 60 και του 70. Να μπορέσουν δηλαδή οι νέοι να αντιμετωπίσουν τον χώρο εργασίας, τον κόσμο της εργασίας που αλλάζει και που εμείς τον χρηματοδοτούμε. In one minute. Μισό λεπτό. Σας δίνουμε να πιείτε λίγο νερό. με συγχωρείτε. Πάντως ε, μπορούμε ε, να, προχωρήσουμε, αν θέλετε, ναι, σε αυτό το διπλό ε, ε παράλληλο δρόμο. και γι' αυτό δεν ήθελα να, να, επικεντρωθώ μόνο σε ένα θέμα. Νομίζω πως απάντησα πάνω κάτω σε όλους. Από τον συνάδελφο που όμως έφυγε, αν κατάλαβα καλά, από την ε, διερμηνία που δεν αμφιβάλλω ε, δεδομένης ε, της ποιότητας της διερμηνίας των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου, Ε, άκουσα μια ολόκληρη σειρά νοησιών και γελίων ε, παρατηρήσεων. Ε, είναι αυτή η αντιευρωπαϊκή ρητορική, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Φαίνονται, φαίνεται τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει, αλλά δεν χρειάζεται να απαντήσω σε τέτοια. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριώτη. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν άλλα ε, σχόλια ή ερωτήσεις από πλευρά σας, ε, σας ευχαριστώ πολύ ε, που ήρθατε εδώ. για αυτήν την ανεπίσημη συζήτηση που μου αρέσουν ιδιαίτερως. Ερωτήσεις, απαντήσεις, διαφωνίες, το χρονοδιάγραμμα υποβολής τροπολογίων είναι 22 Μαΐου. Ε, και στις 19 Ιουνίου θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. και θα μας διευκολύνεται ιδιαίτερως να τα κάνουμε όλα αυτά, μιας και ήρθατε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, νούμερο 7 το οποίο αφορά μία μελέτη σχετικά με την ένταξη των προσφύγων σε Αυστρία, Γερμανία και Σουηδία. Ο συγγραφέας η συγγραφέας της ε, συγκεκριμένης ε, ε μελέτης ε, είναι η κυρία Κον η οποία είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Έρευνας και στη συνέχεια θα σας δώσω το λόγο ε, να ε, θυμάστε ότι ακόμα και αν δεν υπάρχουν αρκετοί στην αίθουσα που παρακολουθούν τη συνεδρίαση, υπάρχουν πάρα πολλοί στα σπίτια από, το, από τους υπολογιστέ τους που μας παρακολουθούν. Ε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω την μελέτη σχετικά με την ένταξη των ε, προσφύγων σε Αυστρία, Σουηδία και Γερμανία ε, ε, που έγινε ύστερα από εντολή της Επιτροπής ΣΥΜΠΛ. Είναι μια συγκριτική μελέτη, οπότε σε 15 λεπτά θα σας πω περισσότερα σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί στις τρεις χώρες όσον αφορά πολιτικές ένταξης και όταν ε, μιλάμε για τις συγκεκριμένες ε, τρεις ε, χώρες, αυτή ήταν οι κύριοι προορισμοί για το 2015 και ως τις αρχές του 2017 για ετούντες ασύλου ασχέτως του πώς εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις ε, χώρες ε, είναι πιο εξελιγμένες όσον αφορά ε, τις παροχές τις παροχές πολιτικών για την ένταξη σε σχέση με την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα υπήρξε μια παρουσίαση παράλληλη έρευνα πριν από ένα μήνα περίπου και όταν ε, βγήκε η συγκεκριμένη έρευνα, οι τρεις χώρες αυτές ήταν λιγότερο προετοιμασμένες ε, στο να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ε, προσφύγων η πολιτική ένταξη λοιπόν ξεκινά σε αυτές τις τρεις χώρες σε αντίθεση ε, με τις ε, τρεις χώρες ε, του Βορρά, Αυστρία, Σουηδία, Γερμανία. Εκεί έχουν πιο ανεπτυγμένες πολιτικές, ιδιαίτερως η Σουηδία για πολλά χρόνια, ενώ η Αυστρία και η Γερμανία εντατικοποίησαν τις προσπάθειες και τους πόρους τους, ιδιαίτερως κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Όταν μιλάμε για αυτό. Πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη σχετικά με την ε, υποδοχή και ένταξη προσφύγων στις τρεις χώρες. Ε, κυρίως ε, καλύπτουμε τα τρία τελευταία χρόνια και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί καθώς επίσης ε, και τις, ε, ε, και προκλήσεις και το περιεχόμενο θα επισέλθω στο ρόλο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης καθώς επίσης και τις αλλαγές αντίληψης στο πολιτικό πεδίο όσον αφορά ε, την ε, ένταξη βασίζεται στην ανάλυση επισήμων εγγράφων καθώς επίσης ε, και ακαδημαϊκών εργασιών όπως επίσης και δεδομένα τα οποία έχουν παραχθεί από την Eurostat καθώς επίσης και από, τα, από τις εθνικές υπηρεσίες. Έχουμε εδώ πληροφορίες σχετικά με τις ροές αναμίνα των ε, ατόμων που κάναν πρώτη φορά αίτηση ασύλου σε Αυστρία, Γερμανία ε, και ε, Σουηδία σε σύγκριση με το πληθυσμό. Το 2015 ήταν υψηλότερο στην Σουηδία ακολούθησε η Αυστρία και η Γερμανία, στη συνέχεια όμως άλλαξε. Ε, υπάρχει έντονη μείωση των ροών μετά τον ε, Μάρτιο του 2016, οπότε και έκλεισε ο, Βελγα... ο Βαλκανικός διάδρομος και είχαμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στην Γερμανία υπήρξε επίσης ε, μία μείωση, η οποία δεν αντικατοπτρίζεται εδώ πέρα στις ε, στατιστικές ασύλου, ε, διότι η Γερμανία έχει ένα σύστημα δύο σταδίων για την αίτηση ασύλου, ε, στην αρχή κάνουν την αίτηση, ε, κάνουν δύο διαφορετικές αιτήσει, το οποίο σημαίνει ότι θα περάσουν αρκετοί ε, μήνες μεταξύ αυτών των δύο σταδίων και τα τελευταία δεδομένα μονάχα του τελευταίου σταδίου δίνονται στην Eurostat. παρόλα αυτά όμως και στη Γερμανία μειώθηκαν οι ροές μετά τον Μάρτιο του 2016 βλέποντας τις πολιτικές ε, ε, ένταξης ε, τα πρώτα χαρακτηριστικά των προσφύγων και των ετούντων ασύλου που έφτασαν τα τελευταία τρία χρόνια στις τρεις αυτές χώρες που κατάγονται από πέντε κυρίως χώρες Συρία η μεγαλύτερη ομάδα Ιράκ, Αφγανιστάν, Ερυθρέα και το Ιράν όμως ε, πρόσφατα κατάγονται επίσης από την Ιγυρία, τη Γεωργία, την Τουρκία, το Πακιστάν. Ο, από αυτές ε, τις εμπόλεμες ζώνες λοιπόν έχουμε ε, κάποια μείωση, πρόκειται κυρίως για νέους, ε, άρενες, το 16 με 17% είναι ε, άνδρες και το 70% είναι κάτω των 30%. Ε, το 20% είναι ασυνόδευτοι ε, που είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα η ηλικία ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο ε, όσον αφορά ε, την εκπαίδευση και όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, το οποίο είναι ένας ε, ένα σημαντικό παράγοντας για την ένταξη ε, στην αγορά εργασίας. Τα οι ε, δεν είναι ξεκάθαρες ακόμα, όμως αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει μια κοινή τάση και στις τρεις χώρες, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος μορφωτικού επίπεδου είναι πολλοποιημένο η πλειοψηφία των Συρίων, Αφγανών και Ιρακινών έχουν τουλάχιστον ανώτερη ε, δευτερεύουσα εκπαίδευση ενώ από τη Σομαλία, Ερυθρέα έχουν ε, ε, τουλάχιστον στην καλύτερη των περιπτώσεων κατώτερη δευτερεύουσα εκπαίδευση και οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν τελειώσει μονάχα την πρωτοβάθμια είναι ε, μια πολύ ε, πολλωμένη εικόνα και όσον αφορά τα ποσοστά αναγνώρισης αυτά είναι αρκετά υψηλά και πάνω από ε, τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 70% στο 16 αναγνωρίστηκε όμως μειώθηκε στο 40 με 50% το 17 Επίσης άλλαξε το είδος ε, της ε, προστασίας που χορηγείται στους ετούντες ασύλου, ένας ε, στους δύο Σουηδία και Γερμανία και ένας στους τρεις στην Αυστρία των επιτυχημένων ετούντων λαμβάνουν επικουρική προστασία και αυτό αφορά ιδιαιτέρως τους Σύριους στην Σουηδία όπου μόλις το 5% των Σύριων ε, λαμβάνει προστασία υπό τη σύμβαση της Γενέβης ενώ το 95% εξ αυτών λαμβάνει μονάχα προσωρινή επικουρική προστασία όλα αυτά έχουν αλλάξει και στην Γερμανία λιγότερο όμως ε, στην Αυστρία δεν υπάρχουν μονάχα ε, όμοια μοτίβα μεταξύ των ε, χωρών αλλά και ε, αντικρουόμενες εξελίξεις, για παράδειγμα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι περιορισμένη η πρόσβαση στην Αυστρία ε, διότι στην ε, Αυστρία τρεις, ε, μετά από τρεις μήνες οι ετούντες ασύλου μπορούν να εργαστούν αλλά μονάχα άδειες εργασίες, άδειες εργασίες δίνονται μονάχα στο πλαίσιο εποχικής εργασίας, στο τουρισμό και στη γεωργία ενώ από την άλλη στην Γερμανία και τη Σουηδία έχει ε, απελευθερωθεί η πρόσβαση στην ε, αγορά εργασίας ε, έχει περιοριστεί η αξιολόγηση για την πρόσβαση εργασίας ενώ στη Σουηδία δίνονται πιο εύκολες οι άδειες εργασίας. Οι ετούντες ασύλου λοιπόν μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται αμέσως αφού υποβάλουν την αίτησή τους ε, υπό ορισμένες ε, συνθήκες χωρίς άδεια εργασίας. Η Αυστρία επίσης ε, έχει ένα χαρακτηριστικό διότι υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε επιδόματα σε ορισμένα κρατήδια της Αυστρίας όμως οι ετούντες ασύλου έχουν πρόσβαση ε, ε, προγράμματα ε, κατώτατου μισθού και αυτό σε αντίθεση με την οδηγία δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοια είναι η αντίδραση ε, στις ε, μεγάλες ε, ροές και στην επιβάρυνση των αρχών για την, για την έγκυρη αξιολόγηση των αιτήσεων και όσον αφορά την, την παροχή δυνατοτήτων φιλοξενίας, διαμονής και οι τρεις χώρες λοιπόν έχουν μια πιο περιοριστική πολιτική ασύλου ήδη πριν από τη συμφωνία με την Τουρκία ε, είχαν εισαχθεί, επανεισαχθεί ε, συνοριακοί έλεγχοι και η νομοθεσία άλλαξε επίσης το είδος ε, της προστασίας με την προσωρινή προστασία να, να γίνεται όλο και πιο, ένα όλο και πιο σύνηθες φαινόμενο στην Σουηδία για παράδειγμα πριν από το 2016 ένας ε, αναγνωρισμένος ε, πρόσφυγας ε, λάμβανε αμέσως άδεια παραμονής, όμως στη συνέχεια παίρνουν μονάχα προσωρινή προστασία. Το ίδιο ισχύει και για την Αυστρία και την Γερμανία, όπου η προσωρινή προστασία μειώθηκε από τα 5 στα 3 έτη αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό και των τριών ε, χωρών. Οι άδειε παραμονής έχουν ε, γίνει, ε, δίνονται με βάση τις μεμονωμένες προσπάθειες ένταξης, όπως για παράδειγμα αν έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων, Ε, και αν ε, προσπαθούν να τα βγάλουν από μόνοι τους ε, πέρα και αυτό έχει γίνει ένα χαρακτηριστικό, ένα νέο χαρακτηριστικό και στις τρεις χώρες. Επίσης το δικαίωμα συμμετοχής σε μαθήματα ένταξης, γλωσσικά μαθήματα για παράδειγμα έχουν γίνει υποχρεωτικά. Οι πρόσφυγες λοιπόν δεν είναι άλλο ε, υποχρεωτικά. Οι πρόσφυγες δεν είναι υποχρεωμένοι ε, να ε, συμμετέχουν σε τέτοια μαθήματα, μπορούν να λαμβάνουν κάρτες επιδομάτων όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση. Είναι κάτι το οποίο συζητάται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα έντονα στην Γερμανία. Ε, είναι κάτι το οποίο όμως συζητάται και στις τρεις χώρες, στην Αυστρία και την Γερμανία. Η λίστα των ασφαλών χωρών προέλευσης έχει επεκταθεί, ενώ από την άλλη η Σουηδία ακόμα δεν έχει μια τέτοια λίστα. ενώ ε, η Γερμανία και η Σουηδία εισήγαγαν ε, περιορισμούς εγκατάστασης για να μπορέσουν να ε, κατανείμουν εισάριθμα την, την κατάσταση σε όλη τη χώρα. Αυτό είχε ως στόχο να μειώσει την ροή των ετούντων ασύλου αλλά και τους παράγοντες που τους προσέλκυαν. Όσον αφορά τις ε, πολιτικές ε, ε, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ε, ενώ ε, ελέγχουμε την, ε, τη διαδικασία ένταξης έχουμε ε, αυξηθεί, έχουν αυξηθεί οι προϋπολογισμοί, η συμμετοχή στην αγορά εργασίας φαίνεται όσο σημαντικότερος παράγοντας υπέρ της μακροπρόθεσμης ένταξης και στις τρεις χώρες και επικεντρώνονται σε αυτό ιδιαίτερος και γι' αυτό το λόγο δίνονται ποσά για την ένταξη στην αγορά εργασίας ε, σε αντίθεση, το οποίο βασίζεται με την έλλειψη εργατικού ε, δυναμικού, ε, ελλείψεις που γίνονται όλο και πιο έντονες και, στις, και πασιφανείς και στις τρεις χώρες. Επίσης, η πολιτική βούληση για αποτελεσματική ένταξη βασίζεται σε μαθήματα και αποτυχίες του παρελθόντος για μια καλύτερη ε, ένταξη στην αγορά εργασία. Οι ε, εργασίας οι ε, παράσχουν πόρους για να ενισχύσουν την ένταξη. Υπάρχει συμφωνία σε βασικά συστατικά στρατηγικών ένταξης ε, υπάρχουν ε, γλωσσικά μαθήματα, συνδυασμό γλωσσικών μαθημάτων με εργασία, ε, επαγγελματική εργασία, εμπειρία. τα οποία θεωρούνται πιο επιτυχημένα και υποσχόμενα υπήρξαν νέες προσεγγίσεις επίσης και νέοι τρόποι για την συμμετοχή των εργοδοτών ε, στην ένταξη και προσοχή στην αξιολόγηση δεξιοτήτων και την αναγνώριση πτυχίων ιδιαιτέρως όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Θα ήθελα να σας δώσω ένα ε, παράδειγμα, η δαπάνη για την ένταξη τριπλασιάστηκε από το 15 στο 17 ε, σε Αυστρία και Γερμανία και αυξήθηκε κατά 10 φορές ε, σε σχέση με τα τελευταία 10 χρόνια στην Σουηδία και το κόστος στην, για τη Σουηδία, για την αξιολόγηση των αιτήσεων, τη φιλοξενία και την διετή υποστήριξη ε, για τα προγράμματα ένταξης αντιστοιχεί με το συνολικό κόστος ε, για ε, την αστυνόμευση και την ανώτερη εκπαίδευση σε όλη την Σουηδία. Αυτό δείχνει πόσο υψηλό είναι το κόστος για την ένταξη παρά την συμφωνία σε βασικά συστατικά των πολιτικών ένταξης υπάρχουν επίσης και εθνικές ε, προσεγγίσεις οι οποίες ποικίλουν λαμβάνοντας υπόψη ε, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συστημάτων αναγνώρισης, ε, πρόσληψης και το πολιτικό κλίμα που επικρατεί για παράδειγμα, αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές όσον αφορά ε, τις, ε, ε, τις επιταχυμένες διαδικασίες ε, στην Σουηδία, ούτως ώστε να απασχοληθούν οι πρόσφυγες, οι υψηλά καταρτισμένοι πρόσφυγες, ενώ σε Αυστρία και Γερμανία επικεντρώνονται στο να γίνεται εκπαίδευση που είναι το, ε, η στάνταρ διαδικασία τα προγράμματα αυτά προσαρμόζονται και σχεδιάζονται έτσι ούτω ώστε οι νέοι σταδιακά να μπορέσουν ε, να ενταχθούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και επίσης έχουμε την πρωτοβουλία 3 συν 2 στην ε, Γερμανία ε, όπου νέοι έως 25 από το Αφγανιστάν για παράδειγμα μπορούν να εισαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα πρακτικής και στη συνέχεια να πάρουν άδεια παραμονής για αυτά τα τρία χρόνια και στη συνέχεια συν δύο χρόνια σε περίπτωση που μπορέσουν να βρουν δουλειά. Υπάρχουν λοιπόν όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες ε, ούτως ώστε ε, οι άνθρωποι αυτοί να συμμετέχουν σε αυτές τις ε, πρακτικές. Ε, η Γερμανία ξεχωρίζει επίσης όσον αφορά την παροχή υποστήριξης ένταξης σε πρώιμο στάδιο όχι μονάχα αφού ε, αναγνωριστούν ως ε, πρόσφυγες, αλλά ακόμα και στη συνέχεια μπορούν να συμμετέχουν σε γλωσσικά μαθήματα, σε προγράμματα ε, απασχολησιμότητας, ε, αλλά αυτό αφορά και αυτούς οι οποίοι έχουν ε, μεγάλη πιθανότητα να παραμείνουν, δηλαδή για άτομα τα οποία κατάγονται από χώρες όπως είναι η Συρία, ή η Ερυθρέα με ε, ποσοστά αναγνώρισης 50% ε, και κάτι άλλο ιδιαίτερο στην ε, Γερμανία είναι ότι το στάτους ανοχής, το καθεστώς ανοχής είναι ένα νομικό καθεστώς. Οι άνθρωποι αυτοί λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό ε, παύσης της απέλασής τους ε, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πηγαίνουν ε, και να συμμετέχουν σε γλωσσικά μαθήματα για παράδειγμα. Αυτό όμως δεν ισχύει στις άλλες ε, χώρες. Τώρα όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας που είναι σημαντική σε αυτές τις χώρες ε, και ό,τι γνωρίζουμε από το παρελθόν. Είναι δύσκολο να, εξ, να αξιολογήσουμε ε, τις συνθήκες εργασίας ε, διότι τα περισσότερα δεδομένα δεν επιτρέπουν να ξεχωρίσουμε μεταξύ ε, των προσφύγων από τους υπόλοιπους ε, μετανάστες όμως το συγκεκριμένο γράφημα που σας παρουσιάζω ε, προέρχεται από το 2014 ε, μια έρευνα για την ε, συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει ότι ένας στους δύο βρήκε μεσοπρόθεσμα εργασία σε σχέση με τους εργατικούς σε σχέση με τους μετανάστευς για λόγους εργασίας ε, και αυτό ιδιαίτερως αφορά τον πρώτο χρόνο το χάσμα τελειώ, ε, ε, κλείνει σε σχέση με τους ντόπιου μετά από 20 χρόνια τα σουηδικά δεδομένα αλλά και τα τελευταία δεδομένα από τη Γερμανία δείχνουν ότι τα ποσοστά αποσχολησιμότητας ελάχιστα ε, βελτιώθηκαν 15% ε, ε, για τον πρώτο χρόνο, 22% μετά από δύο χρόνια σε Αυστρία και Γερμανία και 30% μετά από τρία χρόνια αφού έχουν λάβει καθεστώς ασύλου, ελάχιστα καλύτερα. Όμως γενικά χρειάζεται χρόνο Επίσης, τα εμπόδια για τους πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να μπουν στην αγορά εργασία είναι όμοια με τους ε, μετανάστες ε, ε, είναι διαφορετικά με τους μετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει έχοντας λάβει εργασία και αυτοί είναι και λόγοι για τους οποίους οι ε, πρόσφυγες δυσκολεύονται περισσότερο να μπουν στην αγορά εργασίας. Ε, το ερώτημα τώρα είναι ε, πώς οι πρόσφυγες πρέπει να ενταχθούν στις τοπικές αγορές εργασίας. Αυτό είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Υπολογίζεται γύρω στο 1% της αγοράς εργασίας σε Γερμανία και Αυστρία και γύρω στο 2% στη Σουηδία είναι πολύ γενική υπολογισμοί ε, και για διάφορους λόγους είναι δύσκολο να υπολογιστεί κάτι τέτοιο. όσον αφορά την, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό. Η ένταξη ε, παραμένει ε, στη δικαιοσυνδοσία των ε, κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών από τη μία με ειδικά ταμεία ε, και στη συνέχεια με πιο ε, με συντονιστικά ε, μέτρα, με πρωτοβουλίες κοινή μάθησης, τι γίνεται με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τα κυριότερα ποσά είναι το ε, ΑΜΙΦ, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ε, Ταμείο. Το πρώτο έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαιτέρως, το γνωρίζουμε αυτό από την παράλληλη έρευνα που έγινε σε Ελλάδα, Ιταλία και Ουγγαρία. Σε αυτές τις χώρες επίσης υπάρχει υποστήριξη των, της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, όμως ε, ε, κάτι τέτοιο δεν ισχύει τόσο ε, σε τρεις χώρες το ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρησιμοποιεί τελικότερο για την ε, ένταξη στην αγορά εργασίας, όμως αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια ε, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ESF, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουν μειωθεί οι αρχές διαχειρίζονται τα, τα τα ποσά ε, του ISF δηλώνουν ότι όλα αυτά είναι, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική ε, για παράδειγμα οι αυστριακές υπηρεσίες δεν έχουν υποβάλει αίτηση ε, για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον ESF για αυτή την περίοδο, ενώ στη Γερμανία έχουν μειωθεί. Το ίδιο και στην Σουηδία. οι αρχές ε, δηλώνουν ότι καλωσορίζουν ε, την προσπάθεια ε, για την αύξηση των ποσών που δίνονται για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και έχει γίνει πρόταση από αυτήν την ομάδα σε αυτό το πλαίσιο που τις καλωσορίζουν και οι τρεις χώρες. Όσον αφορά τώρα το ε, πολιτικό κλίμα και το πώς το αντιμετωπίζει ε, ο λαός, ε, εδώ είναι ένα ευαίσθητο θέμα και στις τρεις χώρες αλλά και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι το πιο πιεστικό ζήτημα η συζήτηση γενικά ε, εμφανίζει μεγαλύτερη ε, πόλωση βλέπουμε για παράδειγμα ε, τι λέγεται ε, στις ε, αμερικανικές ειδήσει. Έχουμε αντιμεταναστευτικά κόμματα, όμως ακόμα και στη Σουηδία, παρόλα αυτά όμως η Σουηδία ξεχωρίζει ότι είναι η χώρα όπου σχεδόν το 50% βλέπει θετικά τη μετανάστευση ανθρώπων εκτός της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 20%, στη Γερμανία στο 10% και στην Αυστρία στο 28%. Η Σουηδική κοινωνία υποστηρίζει λοιπόν ιδιαίτερως τους πρόσφυγες και την ένταξή τους και ε, αυτό είναι υψηλότερο. Ε, ε, το ποσοστό κατά της υποστήριξης των προσφύγων είναι υψηλότερο στην Αυστρία. Τώρα όσον αφορά τις προκλήσεις σχετικά με, την, με τις πολιτικές ένταξεις υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον ιδιαίτερος όσον αφορά τις προσωρινές άδειες παραμονής, το οποίο αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα, ούτως ώστε ε, να μπουν σε προγράμματα γλωσσικά και ε, επαγγελματικά ε, το 2016 στην Σουηδία δίνονταν άδειες παραμονής ενώ τώρα μονάχα προσωρινές άδειες παραμονής Το φαινόμενο λοιπόν ότι οι επενδύσεις αποτελούν το ε, κίνητρο, ε, άρα επενδύσεις σε ανθρώπινες δεξιότητες ε, μειώνονται. Επίσης υπάρχουν κενά συντονισμού και στις τρεις χώρες η πολιτική ένταξη αφορά διάφορους τομείς και τμήματα της κυβέρνησης που καθιστούν την ένταξη δύσκολη, η παροχή υπηρεσιών ε, δεν, ε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες απασχόλησης ε, στην Ευρωπαϊκή, στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να παράσουν γλωσσικά μαθήματα, το οποίο δυσχεραίνει το έργο ένταξης και στη Σουηδία ε, οι τρεις βασικές, βασικοί παράγοντες, οι τρεις βασικές αρχές ε, οι ε, κοινότητες, οι ε, υπηρεσίες ένταξης και απασχόλησης ε, θα πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα τρεις διαφορετικές φορές αντί να βασιστούν σε προηγούμενα δεδομένα. Ε, θα πρέπει να δίνεται, να παραχθεί περισσότερη εκπαίδευση και εκπαίδευση ιδιαίτερω ε, σε επαγγέλματα τα οποία ε, ταιριάζουν στις δεξιότητες των προσφύγων αλλά το πρόβλημα είναι ότι πολλοί δεν έχουν βασική εκπαίδευση και υπάρχει λοιπόν ξεκάθαρη ανάγκη μαθημάτων αλφαβητισμού και επίσης ε, χρειάζονται πολιτικές με βάση τις αποδείξεις ε, ε, που θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα με βάση τον προσφυγικό πληθυσμό. Υπάρχουν ακόμα όμως μεγάλες ελλείψεις όσον αφορά τα δεδομένα αυτά Τώρα όσον αφορά τις συστάσεις ε, για τη βελτίωση της ένταξης, της υποστήριξης ένταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να, να θεωρήσουμε ε, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να μειώσουμε το ε, διοικητικό άχθος όσον αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ταμείων Επίσης ε, θα πρέπει να γίνεται χρηματοδότηση ε, βραχυπρόθεσμων ε, και μικρών προγραμμάτων. Θα πρέπει να έχουμε ένα καρουζέλ προγραμμάτων διότι, με αυτό, διότι χάνεται γνώση και εμπειρία. και ε, πέραν από την παροχή χρηματοδότησης για την ένταξη ε, ε, ανέφερα ότι ο βασικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συνεισφέρει στον συντονισμό. Έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο αδράσης για υπηκόους τρίτων χωρών από το 2016 και τα όσα παρατηρούμε εδώ πέρα είναι ότι όταν ε, προωθούμε ε, την ανταλλαγή καλών ε, πρακτικών η ταυτοποίηση των παραγόντων που δημιουργούν εμπόδιο είναι κάτι το οποίο πολλές φορές αγνοείται ιδιαιτέρως από τις δημόσιες αρχές που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα. Τέλος, ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα παρακολούθησης ε, τους δείκτες ε, Σαραγώσα ε, που ε, αφορούν τα άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, το οποίο σημαίνει ε, ότι οι πρόσφυγες δεν αναγνωρίζονται ως ξεχωριστή κατηγορία, κατηγορία στα δεδομένα και θα πρέπει λοιπόν να βρούμε, να βρούμε στοιχεία και καλές πρακτικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν για την συλλογή εμπειρικών δεδομένων. Αυτά λοιπόν όσα ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη που μας παρουσιάσατε. Δεν είναι πολλοί οι ευρωβουλευτές παρόντες, αλλά όποιος έχει ερωτήσεις, παρακαλώ. Η κυρία Ρέτνα από την Αυστρία έχει μια ερώτηση για σας. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για βέλτιστες πρακτικές που θα είχατε να συστήσετε ε, και στους υπόλοιπους. Επίτα, θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για τα κενά συντονισμού. Πρόκειται για τις ικανότητες, ε, σε τι επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας, ε, τι ακριβώς εννοείται. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, ε, δεν χρειάζεται περισσότερη στήριξη για τις γυναίκες πρόσφυγες. Το είπατε, αλλά τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Τι μέτρα προβλέπετε δηλαδή εσείς. Θα ήθελα να μπείτε περισσότερο σε βάθος για αυτά. Εγώ πριν από πολλά βέβαια χρόνια ήμουν σύμβουλος στην Διεθνή Αμνηστία για πρόσφυγες. Πριν από πολλά χρόνια βέβαια, εντάξει, οπότε σίγουρα έχει αλλάξει η κατάσταση πολύ. Αλλά συχνά είχα τότε την εμπειρία όταν έπρεπε να δώσω κάποιες συμβουλές ήταν κυρίως οι άντρες οι οποίοι, οι οποίοι ερχόντουσαν και έλεγαν μάλιστα ότι ερχόντουσαν και εκ μέρους της γυναίκας τους χωρί όμως να έρχεται εκείνη. Οπότε μια σύσταση που θα είχα εγώ να κάνω, αλλά πάλι σα λέω έχει να κάνει με την εμπειρία μου πριν από πολλά χρόνια, ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε απευθεία με του ενδιαφερόμενου. Μπορείτε να μα πείτε περισσότερα και γι' αυτό, αν έχετε επαφή δηλαδή και με γυναίκε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μαρτάν επίση έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Συγχαίρω την κυρία για την παρουσίασή της, που συνήθως είναι 15 λεπτά τέτοιε παρουσιάσεις, αλλά εκείνη την έκανε σε 35. Τέλος πάντων, σε σχέση... Τι να κάνουμε, έτσι καλώς δεν έχουμε πια ευρωβουλευτές εδώ μέσα σχεδόν, οπότε δεν πειράζει που μακρηγορήσατε. Φαίνεται να είναι αντικειμενική και δεν φαίνεται να μεροληπτεί πολιτικά. Θέτεται το ζήτημα εκτός από τη Σοφία, την Σουηδία τέλο πάντων, ότι δεν είναι προφανές το θέμα της υποδοχής των προσφύγων ούτε για τους πρόσφυγες ούτε και για τον τόπιο πληθυσμό. Το είπατε και για τη Γερμανία και το λέτε χωρίς να μεροληπτείτε και σας συγχαίρω για αυτό που επιδείξατε ουδετερότητα στην παρουσίαση αυτής της μελέτης. Ωραία. Για να απαντήσετε τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη για τα 35 λεπτά. Και ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια. Για να απαντήσω τώρα στις ερωτήσεις που έκανε η Ευρωβουλευτής από την Αυστρία, πρακτικά παραδείγματα λέτε, παραδείγματα από την εμπειρία μας. Όπως είπα, ακόμα Υπάρχει θέμα ε, με την γνώση που διαθέτουμε, τι ακριβώς δηλαδή γνωρίζουμε, θετικό ή αρνητικό από την κάθε χώρα. Κυρίως στις βόρειες χώρες που έχουν μεγάλη παράδοση και εμπειρία και προθυμένες πολιτικές, εκεί ξέρουμε τι λειτουργεί με επιδόματα για πρόσφυγες κλπ. Αλλά είναι δύσκολο να δώσω παραδείγματα στην πράξη. Το θέμα της γλώσσας. Να αρχίσει δηλαδή ο πρόσφυγας να μαθαίνει τη γλώσσα του τόπου που διαμένει πολύ γρήγορα. Από την αρχή ε, επαγγελματικής κατάρτισης επίσης μαθήματα βοηθούν πολύ. Έχει φανεί ότι κάνουν τη διαφορά γιατί βοηθούν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες να ενταχθούν έτσι πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Και συνδυάζονται τα γλωσσικά μαθήματα με επαγγελματική εμπειρία. Οπότε αυτό βοηθάει η πρακτική άσκηση, η μαθητεία. σε μια πραγματική επιχείρηση. Είναι κάτι πολλά υποσχόμενο αυτό, σαν παράδειγμα. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, είναι σημαντικό να μάθουμε τι γνωρίζει ο κόσμος, ποια είναι τα προσόντα του. Συχνά δεν έρχονται με επίσημα διπλώματα, έχουν όμως επαγγελματική εμπειρία. Είναι λοιπόν σημαντικό για τις αυστριακές αρχές, αλλά και τις γερμανικές και τις υπόλοιπες, να ξέρουν τι ακριβώς τα άτομα αυτά γνωρίζουν, τι ικανότητες έχουν. Και είναι σημαντικό να γίνεται και η αξιολόγηση και η καταγραφή των ικανοτήτων τους, τόσο των επίσημων, των πιστοποιημένων, όσο και των άτυπων. Η Bundesagentur, που είναι το αντίστοιχο του ΕΔ στη Γερμανία, έχουν ε, εργαλεία πολύ προθυμένα και τώρα θα δοκιμαστούν. Δηλαδή υπάρχουν νέες πρακτικές που τώρα δοκιμάζονται, είναι σε πιλωτικό στάδιο και θα αξιολογηθούν. Ίσως ένα-δύο χρόνια να γνωρίζουμε περισσότερα για τέτοιου είδους πολλαποσχόμενες πρακτικές. Τώρα για τα κενά στο συντονισμό. Υπάρχουν ε, πολλά επίπεδα διακυβέρνησης που εμπλέκονται, οι δήμοι, ε, τα κρατήδια, το ομοσπονδιακό επίπεδο, ε, τα συμβούλια προσφύγων κλπ. Συχνά λοιπόν όντως υπάρχουν κενά συντονισμού. Για παράδειγμα δεν υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων. Έχουν γίνει προσπάθειες να καλυφθούν αυτά τα στις δυναμίες στο συντονισμό στην Αυστρία, όπου υπάρχει κάποια συνεργασία μεταξύ κάποιων αρχών, αλλά παραμένουν ακόμα πολλές τέτοιες αδυναμίες και κενά. Για τις γυναίκες, λέτε περισσότερη στήριξη στις γυναίκες πρόσφυγες. Βεβαίως, έχουμε δει ότι συχνά οι γυναίκες πρόσφυγες έχουν υψηλότερα επίπεδα προσόντων από, από τους άντρες. Παρ' όλα αυτά στην απασχόληση διαπιστώνουμε ότι απασχολούνται λιγότερο και έχουν και λιγότερη επαγγελματική εμπειρία. Ε, προτείνεται να μιλάμε απευθεία με τις γυναίκες. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό πράγματι για να ξεπεράσουμε και τα εμπόδια εξαιτία της νοτροπίας. Στη Σουηδία για παράδειγμα, γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε νέους τρόπους για να απευθυνθούμε στις γυναίκες, έτσι. Οπότε, ναι, στην ε, Σουηδία το προσπαθούμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο κύριος Σούτσε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που μπήκα λίγο καθυστερημένο, όμω ε, υπάρχουν τόσο πολλέ συναντήσει σήμερα, συνεδριάσει. Από αυτά τα οποία άκουσα, νιώθω ότι ζω σε άλλο κόσμο. Είμαι Γερμανός. Από το 2015 στο κρατήδιό μου, στο Ξωνία Άνχαλτ, ε, είχα δει πως είναι η κατάσταση ε, και υπήρχαν πρόσφυγες οι οποίοι δεν φεύγουν επειδή διώκονται ή υπάρχει πόλεμος αλλά ε, επειδή θέλουν να βρουν δουλειά και για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενσωματωθούν. Ε, ένας πρόσφυγας ε, λαμβάνει 600 ώρες ε, γλώσσες και όταν ρωτάμε τους καθηγητές πώς είναι η διάθεση μετά από 2-3 μέρες η κατάσταση είναι τρομακτική. Όταν μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους λένε ότι το έργο μας είναι να βρούμε χρήματα διότι οι οικογένειές μας και εμείς πληρώσαμε χρήματα για να φτάσουμε εδώ και όταν κάνουμε μια άσκηση πρακτική δεν μας επαρκεί χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Οπότε ωραία όλα τα θεωρητικά, όμως ε, ε, από ό,τι κατάλαβα με τα λίγα μου γαλλικά από το συνάδελφο, ε, πιστεύω ότι στη Γερμανία έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, ειδικά με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες, οι οποίοι όμως έχουν δεν έχουν σοβαρούς λόγους όπως ε, ότι διώκονται πολιτικά ή πόλεμο, αλλά ε, ε, φεύγουν για λόγους τους οποίους θα χρησιμοποιούσα και εγώ βέβαια, επειδή θέλουν να βελτιώσουν τις οικονομικές τους συνθήκες. Όμως η κατάσταση στη Γερμανία νιώθω ότι είναι διαφορετική από ό,τι άκουσα, από αυτά τα οποία άκουσα τα τελευταία λεπτά. Ως Σουηδή έχω δύο ερωτήσεις, σχόλια. Κοιτώντας τις εικόνες σας, ε, νιώθω ότι το πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατάσταση. Πρώτον, ε, ελάχιστα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη και δεύτερον, Λίγα από τα ε, τρία κράτη-μέλη έχουν χρησιμοποιήσει τις ε, δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αφορά την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την επένδυση σε ε, διάφορα έργα. Κάτι το οποίο τονίσατε στην εισαγωγή σας τουλάχιστον τρία κράτη-μέλη ε, έχουν κάνει αυτά τα οποία θα έπρεπε και πολλά περισσότερα. Όμως, εφόσον δεν λειτουργεί αρκετά καλά το ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν δύσκολο να έχουμε την πολιτική ε, στήριξη να έχουμε ένα κοινό ε, συμφέρον και δράση και, αυτές, ε, και αυτά τα πλαίσια τα οποία υπάρχουν, όπως είναι για παράδειγμα ε, τα ταμεία έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι όπως θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί. Ε, απλά σας προκαλώ να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ. Ίσως πρώτα ως αντίδραση στο δικό σας σχόλιο για τα ευρωπαϊκά κονδύλια ίσως να ήμουν υπερβολικά και χρησιμοποιούνται αλλά μειώνεται η χρήση τους λόγω του διοικητικού φόρτου θα έλεγα. Ναι, τα κονδύλια είναι σημαντικά. Ξέρω ότι στη Γερμανία είναι σημαντικά και στη Σουηδία που έχω συνομιλήσει με τις αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα κονδύλια και παρόλες τις ε, δυσκολίε και το φόρτο αλλά ήθελα και εγώ να πω ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν καλύτερα αυτά τα κονδύλια. Είναι σημαντικά για την κατάρτιση, την επαγγελματική ή την γλωσσική. Είναι επίση πολύ θετικό και ίσως υπάρχουν παραδείγματα της καλύτερης πρακτικής θα μπορούσαν να, να οργανωθούν καλύτερα βέβαια οι αρμόδιες υπηρεσίες για να απορροφούν καλύτερα και πιο αποδοτικά τα κονδύλια. Τώρα εσείς είπατε ότι ναι, είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία αυτή που ζήσατε και συμφωνώ πως είναι δύσκολο, τίποτα δεν είναι απόλυτα τέλειο. Ούτε στη Γερμανία, ούτε στις υπόλοιπες χώρες. Κάθε άλλο. Έχω και εγώ την προσωπική μου εμπειρία, όπου έχω εργαστεί με ασυνόδευτα ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Έχουν τόσο, ε, φαίνεται να έχουν τόσο μεγάλο κίνητρο να μπουν στην κοινωνία, να βρουν δουλειά. Δεν έχω δει ποτέ τόσο ε, πρόθυμους ανθρώπους Είναι δύσκολο να πούμε αυτή η μεικτή μετανάστευση, δηλαδή για οικονομικούς ε, λόγους ή ε, η, προσφυγική, η προσφυγική λόγω πολέμου, συχνά είναι δύσκολο να κάνουμε τη διάκριση. Συμφωνώ μαζί σας ότι πολλοί ότι στη Γερμανία το στάνταρ η στάνταρ πορεία της επαγγελματικης καταρτισης κατάρτισης είναι δύσκολη γιατί διερκεί δύο-τρία χρόνια. Είναι δύσκολο να πείσει τους νέους να το ακολουθήσουν και παίρνουν λιγότερα χρήματα αμείβονται λιγότερα χρήματα. Ενώ αν ξεκινήσουν μια ανεδίκευτη ε, θέση, Αμέσω αρχίζουν να κερδίζουν χρήματα και πρέπει να στείλουν χρήματα πίσω στην οικογένεια που έχει μείνει πίσω. Αν δούμε όμως τα νούμερα, βελτιώνεται η κατάσταση. Όλα και περισσότεροι νέοι αρχίζουν ε, διπλή κατάρτιση. Νομίζω πως οι εργοδότες έχουν να παίξουν ένα μεγάλο ρόλο εδώ, να πείσουν δηλαδή τους ε, πρόσφυγες να ακολουθήσουν και μια μαθητεία. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή και είμαι βέβαια ότι θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον. να δούμε πώς ε, εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ε, πολλά, πολλές προτάσεις, ενδιαφέρουσες προτάσεις, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα συν το χρόνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε, που μας κάνατε αυτή την εισήγηση και που μας αφήνετε και μια περίληψη ώστε να το μελετήσουμε και μόνοι μας. Η μελέτη λοιπόν βρίσκεται εκεί πίσω στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και έχουμε το σημείο 8 στις ενημερίσια διάταξη που είναι τα διάφορα. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα, οπότε κλείνουμε εδώ τη συνεδρίασή μας και στις 2 ακριβώς λέει η Πρόεδρος, θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ να είστε στην ώρα σας για τις ψηφοφορίες. Στην ημερήσια διάταξη λέει 2.30 πάντω. Α, συγγνώμη, 2.30 είναι. 2.30 θα ξεκινήσουμε. τι ψηφοφορίε. όχι στι 2, έκανα λάθο. 2.30.